Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο τμήμα τη σημερινή μα συνεδρίασης και είμαστε στο σημείο 8. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική με τον κύριο Μάρο Σεύκοβιτ, Αντιπρόεδρο Αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση και έχουμε και την κυρία Ελισπιέτα Μπιένκοφσκα, που είναι επίτροπο αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Τώρα στην αρχή πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που είσαστε εδώ μαζί μας. Αυτή τη φορά είναι κάπως ασυνήθιστο το θέμα. Και συμφωνήσαμε ότι κάποιες ερωτήσεις που δεν είναι ακριβώς για αυτό το θέμα θα μπορούσαν να τεθούν και στους δυο σας. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί δεν θα έχουμε την δυνατότητα να συναντηθούμε μαζί σας πια παρά μόνο τον Ιανουάριο ή και τον Φεβρουάριο μάλιστα. Επειδή αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο, αν δέχεστε, οι συνάδελφοι, μια-δυο ερωτήσεις μπορούν να τις υποβάλουν για άλλα ζητήματα πέραν αυτών. Η Ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής μας με τους Επιτρόπους λαμβάνει χώρα τακτικά, ακριβώς στα πλαίσια αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου, όπως είπα πριν. 26 Οκτωβρίου, για παράδειγμα, ε, δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις προκλήσεις ενός κλάδου που εξελίσσεται συνεχώς και αλλάζει συνεχώς και για να κρατήσει μία ηγετική θέση. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι και αύριο θα συζητήσουμε για τη στρατηγική. Συνεπώς, κύριε Αντιπρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί Μιακόφσκα. Είναι μεγάλη χαρά που μπορώ και βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική, την οποία η Κομισιόν υιοθέτησε πριν από μικροχρονικό διάστημα. Πρόκειται για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ξέρω ότι πολλοί εδώ στην Επιτροπή σας παρακολουθούν τη διαστημική ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία χρόνια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στο χώρο του διαστήματος και οικονομικά και πολιτικά και στρατηγικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη στήριξή σας σε αυτήν τη διαστημική μας πολιτική και θέλω να περάσω το μήνυμα ότι είναι ξεκάθαρο πως το διάστημα είναι ο χώρος εκεί όπου η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί. Όπως γνωρίζετε, το διάστημα είναι ένας χώρος ο οποίος κάνει την φαντασία μας να καλπάζει. Όλοι όμως ξέρουμε ότι δεν φτάνει να ονειρεύεται κανείς. Και είμαστε εδώ ώστε τις δυνατότητες που έχει το διάστημα να τις θέσουμε στην υπηρεσία της Ευρώπης και των πολιτών της γιατί το διάστημα και ο διαστημικός κλάδος αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά πολλών τεχνολογιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την οικονομία μας, την ασφάλειά μας, τις μεταφορές μας, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε το 21% του συνολικού κλάδου του διαστήματος, με εκατομμύρια ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, επιχειρήσεις, που έχουν το 1 τρίτο της συνολικής αγοράς και η Ευρώπη έχει μεγάλο μερίδιο στις εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα. Ένα μέρος του ΕΠ εξαρτάται από τις τεχνολογίες του διαστήματος και γίνεται όλο και περισσότερο. Πολλοί οικονομικοί κλάδοι εξαρτώνται από τις δυνατότητες παρακολούθησης από το διάστημα. Ε, είναι εφαρμογέ που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα και στα αυτοκίνητα, στα αυτόνομα αυτοκίνητα που οδηγούνται χωρίς οδηγό. Γιατί λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη αποτελεί σημαντικό παίκτη. Είμαστε και πελάτης, είτε για τους δορυφόρους, είτε γενικότερα για τεχνολογία και 12 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2014 με το 2020 θα έχουμε δαπανίσει στα ερευνητικά μας προγράμματα σε αυτό το τομέα. Είμαστε ο πιο σημαντικός πελάτης του κλάδου και συνεισφέρουμε σε πολλά έσοδα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε όλα αυτά και να ενισχύσουμε το ρόλο μας ακόμη περισσότερο στρατηγικά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κοινέ προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, και να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή αυτονομία όπως επίσης να φέρουμε και αποτελέσματα στις διάφορες πολιτικές μας προτεραιότητες, ασφάλεια, κλίμα, μεταφορές, ε, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κλπ. Γιατί πρέπει να δράσουμε τώρα. Γιατί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο δεν είναι δεδομένη. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο κλάδος. Όλο και περισσότερες χώρες η Κίνα και η Ινδία, για παράδειγμα, δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος. Εδώ μάλιστα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και νέες τεχνολογίες για δορυφόρους ε, και βλέπουμε να γίνονται εκτοξεύσεις και από άλλες χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε καταρτισμένοι και εδώ στην Ευρώπη και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα προσόντα να παραμείνουν στην Ευρώπη. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία τώρα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Στρατηγικής και τι είναι νέο στο έγγραφο το οποίο σας παρουσιάζουμε. Η συνάδελφος θα σας παρουσιάσει σε λίγο τα της στρατηγικής πιο συγκεκριμένα, κυρία Μπιακόφσκα. Επιτρέψτε μου εμένα να σας πω πράγματα που έχουν να κάνουν με το κόστος. Δεν ε, υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική αυτή αν δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε και αν δεν μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος. Αυτοί οι οποίοι έχουν καταφέρει να μειώσουν το κόστος θα έχουν νέες ευκαιρίες στο μέλλον. Το είπε και ο ίδιος Ομπάμα πριν από μερικούς μήνες. Μέρος της στρατηγικής αυτής λοιπόν είναι να προχωρήσουμε τα διαστημικά μας προγράμματα και 30 δορυφόρους να στείλουμε στο διάστημα μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει και μια προβλεψιμότητα για τον κλάδο και περιορισμό των δαπανών για μας. Έτσι το Vega e ή το Arian 6 θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Οι χώρες μέλη συμφώνησαν και για το ΆΡΙΑΝ 6 στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος από ό,τι άκουσα. Και αυτό βέβαια είναι κάτι θετικό. Πρέπει να επικεντρώσουμε λοιπόν την έρευνά μας και την καινοτομία μας στις νέες τεχνολογίες εκτόξευσης δορυφόρων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογίες του διαστήματος του αύριο θα γίνουν κτήμα μας, αντί να μένουμε πίσω. Δεύτερον, η στρατηγική εξετάζει και την θέση την ανταγωνιστική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του κλάδου. Σημαίνει ότι ο Γαλιλαίος πρέπει να επεκταθεί πλήρως και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί. Αυτό βοηθάει την κινητικότητα για το μέλλον, πολλούς τομείς δηλαδή και πολλές υποδομές. Χρειάζεται πρόσβαση επίσης στην τεχνολογία καθοδήγηση από δορυφόρο, κάτι το οποίο χρησιμοποιούν οι τρίτες χώρες. Στα πλαίσια αυτά οι τέσσερι δορυφόροι Γαλιλαίο από τη Γαλλική Γουιάννα που θα εκτοξευθούν όπου να είναι και το Αριάννα 5 αποτελούν στοιχεία κλειδί. Στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών επίσης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών έχουμε τον Κοπέρνικο και το διάστημα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ προκειμένου να πετύχουμε φύ τρόπο τους στόχους μας για προστασία του κλίματος. Επίσης υπάρχουν εφαρμογές και στην ασφάλεια θα σπεί περισσότερα η Επίτροπος Μιακόφσκα. Όλοι αυτοί οι στόχοι απαιτούν κοινέ προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος αποτελεί ένα χωριστό οργανισμό και ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας να προχωρήσουμε στην διαδικασία που ακολουθεί η υπηρεσία αυτή. Η υπηρεσία αυτή λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χωριστούς ε, ρόλους μεταξύ τους, αλλά πρέπει να συνεργάζονται. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και επιβεβαιώθηκε αυτό το πνεύμα συνεργασίας στην κοινή δήλωση που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες όσον αφορά τους στόχους της Ευρώπης για το διάστημα. Βέβαια, απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και των κλάδων. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, με όλες τις λεπτομέρειες τη στρατηγική αυτή και να διευκρινίσει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή. Αυτό ισχύει για την νομοθεσία που πρέπει να προετοιμάσουμε, αλλά και για τη δημοσιονομική στήριξη που θα χρειαστεί η στρατηγική. Χρειάζεται συνέχεια για τα εμβληματικά μα προγράμματα για το 2020, για τα ερευνητικά μα προγράμματα και χρειαζόμαστε και δημοσιονομική στήριξη για να αντιμετωπίσουμε τι νέε προκλήσει κλιματική αλλαγή και ό,τι άλλο είναι στου στόχου μα. Όλα αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζονται λοιπόν στι επόμενε ε, πολιτικές δημοσιονομικέ προοπτικέ. Τώρα, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στην συνάδελφο κυρία Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητέ Μάρος. Ασυνήθιστο θέμα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, νομίζω ότι με την υποστήριξή σας και με την κοινή δουλειά με τον Μάρος ε, θα είναι μόνιμο θέμα συζητήσεων του Κοινοβούλιο, όπως είπε ο Μάρος. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα ε, μέλλοντος τραφές και πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα θυμόσαστε ότι πέρσι Είχα πει ότι έχουμε δύο στόχους για τη δράση μας στον τομέα της διαστημικής πολιτικής το 2016. Ένα στόχος ήταν να επιταχύνουμε την εκτόξευση των δορυφόρων του Γαλιλαίου, του συστήματος Γαλιλαίος, με έξι δορυφόρους φέτος. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι τέσσερις νέοι δορυφόροι ε, εκτοξεύτηκαν στις 17, θα εκτοξευτούν 17 Νοεμβρίου και θέλουμε να υφετήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το διάστημα φέτος Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος και είμαι υπερήφανη που εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τον Μάρος και έχει προχωρήσει τώρα. Από τις 26 Οκτωβρίου είχαμε θετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αδιαστημική πολιτική. Είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό, διότι είναι η πρώτη φορά που υθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τέτοια πλήρη κοινή προσέγγιση και όραμα για τις μελλοντικέ διαστημικές μας ε, δράσεις. Όπως μας είπε και ο Μάρος, κινηθήκαμε στην υπογραφή και το λέω τώρα αμέσως γιατί θα αναφερθώ και στους λόγους τους οποίους ε, η στρατηγική προωθείται και τι περιέχει. Όπως έλεγα λοιπόν, ξεκινά με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Είναι πολύ σημαντικό διότι δείχνουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Έχουμε κάπως διαφορετικούς στόχους με την ΕΖΑ, αλλά όλοι συνεργαζόμαστε και έχουμε δημιουργήσει πολύ ισχυρούς δεσμούς την τελευταία δεκαετία ε, διότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι ο βασικός μας εταίρος όσον αφορά τα δύο βασικά μας προγράμματα, το Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Θέλουμε να πούμε για την ώρα, είναι η δεύτερη διαστημική δύναμη στον κόσμο η Ευρώπη και για την ώρα μπορούμε να υπερηφανευόμεθα για τα επιτεύγματά μας Βέβαια οι προκλήσεις μας αναμένουν και αυτή η στρατηγική νομίζω έρχεται μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ε, και το Γαλιλαίος και το Κοπέρνικος ξεκινούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν και θα λειτουργούν και θα παράξουν ε, στοιχεία για να πει ακριβής η ανάπτυξη των υποδομών του Γαλιλαίος ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση και οι προεργασίες που θα παρέχει το Γαλιλαίος θα ξεκινήσουν και θα έχουμε πλήρη δυναμικότητα το 2020 όσον αφορά το Γαλιλαίος και οι υπηρεσίες του Κοπέρνικου ήδη λειτουργούν μέσω των πρώτων τεσσάρων δορυφόρων. Άλλοι τρεις δορυφόροι θα εκτοξευθούν του χρόνου και άλλοι δύο δορυφόροι μέχρι το 2021. Άρα έχουμε δύο πλήρες συστοιχίες τα επόμενα δορυφόρων. Είναι καμπή, κομβικό σημείο στην στη μας στρατηγική. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε την προσοχή μας από τις υποδομές και δημιουργία υποδομών στη συγκεκριμένη εφαρμογή και υπηρεσίες που θα βασίζονται σε διαστημικά δεδομένα. Πρέπει να οργανώσουμε την απόσβεση των επενδύσεων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι η μόνη ε, διαστημική δύναμη που εστιάζεται επί της ε, ε, πτυχής της αγοράς όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα. Ο διαστημικός τομέας βέβαια ε, μεταμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε νέους ανταγωνιστές, νέες τεχνολογίες, ε, νέα μοντέλα επιχειρηματικά ε, και πολλά μεγάλα, πολύ μεγάλα κεφάλαια κινδυνού και έχουμε πολλές εταιρείες που είναι στην πρώτη γραμμή, ε, ευρωπαϊκές εταιρείες, σοφά τις ξεφτές εκτοξευτές κλπ. Ποιοι είναι οι στόχοι μα όσον αφορά τη συστημική πολιτική, θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη του διαστήματο για την κοινωνία και την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όπω προανέφερα, δημιουργώντα μια ευρωπαϊκή αγορά για εφαρμογέ που βασίζονται στο διάστημα και υπηρεσίε παρόμοιε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα Γαλιλαίο θα χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητά μα, στα τηλέφωνά μα και θα προστατεύει και σημαντικέ υποδομέ κρίσιμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα στοιχεία του Κοπέρνικο, κυρίω για νεοειφεί επιχειρήσει ξεκινώντας ε, τις πλατφόρμες που θα βασίζονται στη βιομηχανία και θέλουμε τα εργαλεία τα διαστημικά να χρησιμοποιούνται καλύτερα μέσω προτεραιοτήτων, α πούμε, αντιμετώπιση αλλαγή του κλίματο, μετανάστευση, άμυνα, κινητικότητα, διασυνδεσιμότητα, ψηφιακή οικονομία κλπ. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα, διότι η Ευρώπη και η διαστημική τη βιομηχανία θα πρέπει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή στον αφορά την καινοτομία. Η δημόσια χρηματοδότηση, ξανά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, θα παραμείνει σε κεντρικό επίπεδο και αυτό το κοινοβούλιο και οι συζητήσεις μας είναι κρισίμου σημασία από αυτή την πλευρά. Θα πρέπει να προωθήσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και επιμερισμό του κινδύνου πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Αυτό απαιτεί πραγματικά αλλαγή νοοτροπίας αλλά αυτό συμβαίνει σε άλλα μέλη του, μέρη του κόσμου, οπότε θα μπορούσε να συμβεί βέβαια και στην Ευρώπη. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε την ανάδυση δυναμικών ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων για διαστημικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα υποστηρίξουμε τη χρηματοδότηση αυτών των διαστημικών νεοφυών επιχειρήσεων. Θέλουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το μελλοντικό αυτό πανευρωπαϊκό ταμείο για τα ταμεία να υποστηρίξουμε τις νεοφύς επιχειρήσεις στον τομέα και να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις. Βασικό κλειδί για τις νεοφύς επιχειρήσεις να εξασφαλίζουμε μια πρώτη σύμβαση για αυτές. Αυτό είναι κάτι που λειτουργεί άριστα στις ΗΠΑ με πολλές νεοφύς επιχειρήσεις που συνδέονται με συμβάσεις της ΝΑΣΑ. Πρέπει να δούμε πώς στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία μπορούμε να προωθήσουμε μια προσέγγιση σύναψης πρώτης συμβάσεως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του διαστήματος. Επόμενο, ε, είναι στρατηγικό στοιχείο σημαντικό το διάστημα και κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στατικής Αυτονομίας. Είναι από τα βασικά ταμπού που καταρρύπτουμε. Θέλουμε όμως να ενισχύσουμε τη συλλογική άμυνα και ασφάλεια και είναι βασικό κλειδί για αυτά οι διαστημικές τεχνολογίες για να έχουμε μια αντοχή και αυτονομία, να μπορούμε να δράσουμε. Εδώ ε, απηχούμε την έκθεση του Κοινοβουλίου που συνέταξε ο κύριος Ντροζιεύσκη με τον κύριο Μαρινέσκου ε, από αυτή την Επιτροπή. Ε, από αυτή την έποψη η στατική που θα ενισχύσει τη διτή χρήση του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικος και το παρόν σύστημα ανείχνευσης, ηχνηλάτησης ε, στο διαστημικό θα εξελιχθεί πλήρως σε, σε ένα σύστημα εντοπισμού ευρωπαϊκό, διαστημικό σύστημα και θέλουμε να δημιουργήσουμε και το GovSatcom, μια πρωτοβουλία για κυβερνητικής χρήσεως δορυφόρους επικοινωνιών. Είναι κάτι απαραίτητο για ανθρωπιστικές κρίσεις, για κατεπίγουσα ανάγκη, εποπτεία των συνόρων και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Ε, όμως αυτή η φιλόδοξη στρατηγική δεν θα ήταν εφικτή χωρίς μια αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εκτοξευτήρων που θα είναι αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος, αξιόπιστη και ανταγωνιστική. Αριάν 6 και Vega C είναι αυτοί οι εκτοξευτήρες. Είναι κρίσιμο για την Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαίτερω που τα, τα μελη τη ΕΣΑ συμφώνησαν όσον αφορά του μηχανισμού εκτόξευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να ομαδοποιήσει τι υπηρεσίε εκτόξευση στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να λειτουργήσει σαν ευφυή πελάτη στον το πρόγραμμα αυτό. Κλείνοντα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κάτι που πιστεύω ότι είναι και ο Μάριος και εγώ ότι είναι μια φιλόδοξη στρατηγική για το διάστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ φιλόδοξα πρόγραμμα. πολλαπλώ ανταποκρίνεται σε θέσει και τίματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρονται σε διάφορε εκθέσει, αλλά και στι συζητήσει μα. Ελπίζουμε, συνεπώ, ότι θα μοιραστείτε αυτή την άποψη και θα υποστηρίξετε αυτή τη φιλοδοξία και τη φιλόδοξη στρατηγική. Ε, γνωρίζουμε ότι η φιλόδοξη διαστημική στρατηγική είναι κάτι που απαιτεί και φιλόδοξα και επαρκή μέσα. Κλείνοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι το διάστημα είναι συγκεκριμένο και θετικό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί στην Ευρώπη. Καμία ευρωπαϊκή χώρα από μόνη τη, κανένα κάτω μέσα από μόνο του μπορεί να τα πετύχει αυτά. Είναι ένα παράδειγμα μια Ευρώπη που λειτουργεί και μπορούμε να συνεργαστούμε. Γι' αυτό είμαι πεισμένη ότι μαζί μπορούμε αυτή την στατική μας να μετατρέψουμε σε μια ομαδική επιτυχία της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους για τις θαυμάσιες παρουσιάσεις τους που είναι πολύ χρήσιμες για όλους μας. και ξέρετε ότι είναι μια καινούργια ιδέα η στρατηγική για το διάστημα. Είναι μια καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και δεκαετίες είναι αυτό το οποίο δεν είχε γίνει και είναι μια πολύ καλή ιδέα για να προωθήσουμε την περιττέρω ολοκλήρωση για το θέμα αυτό. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Οι συντονιστές και οι αντικαταστάτες τους από το, από το ΕΛΚ, ο κύριος Πολ Ρούμπικ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση καταδεικνύει πλήρως ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει μια θετική αντιμετώπιση <clears throat> για τα θέματα του διαστήματος και η διαστημική πολιτική είναι ένα cornerstone, είναι ένας ακρογωνίος λίθος της ε, προσπάθειας αυτής. Θέλω να συγχαρώ τους δύο επιτρόπους, γιατί αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα εν ώψη του μέλλοντος. Στις 16 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, η ΣΤΟΑ θα έχει μια συζήτηση και για την διαστημική πολιτική. Είναι η ετήσια εκδήλωση που γίνεται από την ΣΤΟΑ και νομίζω ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια και στον τομέα των επιστημονικό να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, να <clears throat> έχουμε περισσότερη ανταλλαγή ε, απόψεων μεταξύ επιστημόνων για το πώς ο πληθυσμός της γης που θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια το 2025 να μπορεί να διακινείται και το ίδιο να ισχύει και για τα δεδομένα. Επίσης μας ενδιαφέρει η ύπαρξη βιωσίμων πόρων. Θα είμαστε δέκαδες εκατομμύρια άνθρωποι και είναι όλο και περισσότερο σημαντικό τα τελευταία χρόνια η, η απεικόνηση του πραγματικού κόσμου του πραγματικού κόσμου στον εικονικό κόσμο με τους νέους αλγορίθμους και τις διαδικασίες που έχουμε αναπτύξει και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα πρέπει όσο δυνατόν ταχύτερο να επιτύχουμε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Θα ήθελα επίσης να, σκεφτώ πώς, να, να μάθω πώς η Κομισιόν σκέφτεται να δημιουργήσει την απαραίτητη επικοινωνία για τα θέματα αυτά. Η ΣΤΟΑ έχει πάντα το, το μέλημα να ξεπεράσει τα στεγανά στην επικοινωνία, γιατί κάθε φορά λέμε έχουμε τον α, β, γ, δ τομέα, αλλά Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Υπάρχει καλή διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα και έχετε κάνει κάποια προσπάθεια να δείτε <clears throat> πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ όλων αυτών των φορέων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και είναι απαραίτητο να μπορέσει να γίνει μια μεγαλύτερη διασύνδεση της ψηφιακής πολιτικής μας και της πολιτικής ηλεκτροκίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαστημική πολιτική. Επίσης, στον τομέα της νανοτεχνολογίας γίνονται πολύ σημαντικές πρόοδοι και εδώ θα προκύψουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα ε, υπολογιστών και να εξασφαλίσουμε και την ουδετερότητα αυτών των δικτύων. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα λοιπόν για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των δικτύων. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια σημαντική ενέργεια, ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διευρύνετε τα σύνορα της γνώσης και της τεχνογνωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε να έχουμε αύριο μια ευρύτερη εικόνα της αγοράς για όλα αυτά τα προϊόντα και μια καλύτερη αντιμετώπιση αυτής τη αγοράς. Ο κύριος Σταντίκα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο να, χαρά, να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Σεφτσοβιτς και της κυρίας Μπιανκόφσκα. Είναι μια μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ και σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, δεδομένου ότι έχουμε ενώπιον μας ένα τομέα όπου κατανοούν όλοι την σημασία που μπορεί να προκύψει από μια συνεκτική πολιτική στα διαστημικά θέματα για την Ευρώπη. Στην Επιτροπή μας μιλάμε πολύ για πράγματα που είναι λιγότερο δυσνόητα, όπως είναι η εμπορία εκπομπών, που ενδεχομένως έχει και μεγαλύτερη επίπτωση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά η διαστημική στρατηγική φαίνει με ορισμένα νέα στοιχεία που πρέπει να τα υπογραμμίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια ισχυρή στρατηγική διαστήματος και χωρίς μια σημαντική παρουσία στην εξερεύνηση του διαστήματος. Είτε υπάρχει κανείς σε αυτό το τομέα, είτε δεν υπάρχει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλτ Τραμπ προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη να τα βγάλει πέρα μόνη τους βέβαια, μιλούσε ο Τραμπ για τον στρατιωτικό τομέα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και η διαστημιακή πολιτική είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσετε κάτι το οποίο νομίζω ότι θα βελτιώσει και την υποστήριξη από όλους τους ε, πολίτες μας. Θα πούνε 12 δισεκατομμύρια. Πολύ καλός. Αλλά τι θα προκύψει από αυτά. Να υπάρχει λοιπόν μια καλύτερη επικοινωνία από την πλευρά της Κομισιόν για τα θέματα αυτά θα είναι ένα μεγάλο πλέον έκτημα. Τι θα προκύψει λοιπόν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ως όφελος. Αναφέρθηκα σε ορισμένα από αυτά. <clears throat> Αλλά θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα πώς θα αποκομίσουν ωφέλη τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα από όλα αυτά. Και ποιες θα είναι οι πρακτικές εφαρμογές οι οποίες θα αναπτυχθούν με αυτές τις ενέργειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα φέρουμε προς θεμενή αξία, πώς θα υποφεληθούμε από αυτή τη νέα τεχνολογία με την παρουσία μας στην στο διαστημικό χώρο και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες και αυτές, τι τεχνολογίε, τις τεχνολογίες που θα είναι προ όφελο του Ευρωπαίου πολίτη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και το κάνουμε σε σαφέ στου πολίτε μα, θα έχουμε μεγάλη υποστήριξη από αυτού. Ο τρόπο επίση με τον οποίο θα χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από την επιτυχία τη επικοινωνία. Όλοι προσέχουν αυτά τα οποία λέμε και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία ως στοιχείο αυτής της συνολικής στρατηγικής. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για τις παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος από το ECR, ο κ. Στασανόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία της Κομισιόν που παρουσιάστηκε από του επιτρόπου Μπιενκόφσκα και Σεφτσόβιτ. <clears throat> Χαίρομαι για το γεγονό ότι ήρθατε και οι δύο ομού στην Επιτροπή μα, Αυτό μου δείχνει εμένα ότι αποδίδεται μια μεγάλη σημασία στη διαστημική μηχανία. Και επίσης θέλω να σας συγχαρώ για την στρατηγική διαστήματος που έχετε παρουσιάσει και η οποία έχει μόλις εγκριθεί, διότι πιστεύω ότι καταδεικνύει με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Εμείς έχουμε προετοιμάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με τα θέματα αυτά πρόσφατα και πολλά από τα σημεία τα οποία είχαμε υπογραμμίσει εμείς περιλαμβάνονται και στη στρατηγική διαστήματος της Κομισιόν. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτού του σύνολου τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος και ε, των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν για τη βιομηχανία. Είναι καιρός λοιπόν να υποστηριχθεί αυτή η στρατηγική και ο κλάδος του διαστήματος και χρειάζεται ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα είναι φιλόδοξο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό που μας δίνει ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος για τα νέα συστήματα τα οποία θα εξελιχθούν στο μέλλον και πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών ε, συσκευών και κυκλωμάτων που θα μπορούν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που θα μας δίνει ο Γαλιλαίος. Έχουμε ορισμένα ερωτηματικά βέβαια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα το GOSATSCOM μπορεί και αυτό το πρόγραμμα να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Και ένα ερώτημα για τον Επίτσα Εύτσοβιτς για τη μελλοντική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένα συνεργός συμμετέχων και έχει δώσει μεγάλη ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα αυτά της διαστημικής τεχνολογίας. Ήταν σημαντική και η χρηματοδοτική του συμμετοχή, έχει παράσχει υποδομές στο πρόγραμμα αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπογραμμίσω περισσότερο την σημασία του να υπάρχει διασύνδεση όλων των συστημάτων που αναπτύσσονται. Αλλά βέβαια γνωρίζω ότι δεν έχει εκτοξευθεί ή υπήν το Brexit ακόμα. Αλλά υπάρχει φόβος να αποχωριστούν μεταξύ τους οι δύο πλευρές. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, τονίζω, να υποστηχθεί η συνεργασία στον κεφαλαιόδη αυτό τομέα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ για ένα τόσο νευραλικό τομέα να μην έχουμε τον σημαντικό αυτό εταίρο ο οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα την εταιρική μα σχέση. Θα ήθελα αυτή η εταιρική σχέση να γίνει και πιο στενή. από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι. Ευχαριστώ πολύ για το όσα μας είπατε. Μπορώ να αρχίσω με συγχαρητήρια για το έργο σας όσον αφορά την στρατηγική αυτή του διαστήματος. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα που έχουμε συζητήσει τους τελευταίους μήνες εδώ, πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε τη συμμετοχή, την ενεργό και έντονη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το υπογραμμίζουμε αυτό. Θέλουμε καλύτερη διασύνδεση με την ε, πρωτογενή οικονομία. Θέλουμε και τα στοιχεία για την πλατφόρμα διάδοσης των δεδομένων και πρόκειται επίσης και για αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Είναι πράγματα αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Αλλά, πάντα υπάρχει αλλά, παρόλο που υπάρχει μεγάλη ισορροπία, δεν είναι πολύ ελκυστικό το έγγραφο αυτό. Και γιατί λέω ότι πρέπει να είναι ελκυστικό, δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά γιατί αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, πρέπει να αρέσει στον κόσμο. Και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε πολλές συζητήσεις για παντός είδους επενδύσεις, επενδύσεις σε υποδομές, αλλά 9 στις 10 φορές πρόκειται για επενδύσεις σε παραδοσιακές υποδομές, σε δρόμους, σε σιδηροδρόμους. Αν είμαστε τυχεροί, η Επιτροπή μας αυτή προτείνει και επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, και σε οπτικές ίνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι θα κάνετε και εμεί θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να δημιουργήσετε περισσότερη συνειδητοποίηση όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο γενικό κοινό ώστε να καταλάβουν όλοι πόσο μεγάλη σημασία έχει το διάστημα στην καθημερινή μας ζωή είτε πρόκειται για τα GPS, είτε πρόκειται για τη συνδεσιμότητα είτε για οτιδήποτε άλλο. Μερικές φορές καταλαβαίνουμε ότι οι δορυφόροι είναι σημαντικοί για τη γεωργία. Για παράδειγμα, είναι ένα μόνο παράδειγμα εφαρμογής που μπορούμε να έχουμε με πληροφορίες που παίρνουμε από τους δορυφόρους. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να υπάρξει συνδυτοποίηση πάνω σε αυτό. Και μια ερώτηση κάπως πιο λεπτομερή. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τις ε, πλατφόρμες υπηρεσιών που προσφέρουν ε, πρόσβαση σε δεδομένα παρατήρησης της γης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα προχωρήσει, θα ελοπίσει αυτό το σχέδιο. ώστε με την πλατφόρμα αυτή να έχουμε περισσότερο ωφέλη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Αντιπρόεδρος Χογίψη. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχω μερικές παρατηρήσεις, λέει ο κύριος Είναι πολύ ωραίο να έχουμε νέους εκτοξευστές, Αριάν 6 κλπ. Αλλά έχω και μια ερώτηση. Για τους εκτοξευτές αυτούς θα έχουμε και νέα καύσιμα, γιατί τα παραδοσιακά καύσιμα, τα συμβατικά, δεν είναι καλά για το περιβάλλον. Και έχουμε ακούσει από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ετοιμάζουν τέτοια οικολογικά καύσιμα για εκτοξευτέ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο και για μας αυτό, για τους δορυφόρους μας και για να μπορούμε να προβαίνουμε σε συγκεκριμένε δράσεις, να μπορούμε να διαβάσουμε τα νούμερα στις πλάκες των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, από δορυφόρους παραδόσεις επίσης θα είναι πιο εύκολο. Θα μπορούμε να εντοπίσουμε υγρασία ή άλλα στοιχεία της γεωργικής παραγωγής. Θα βοηθούσε δηλαδή σε πολλά και στο ναυτικό, στις ε, μεταφορές στη θάλασσα. Θα βοηθούσε την αλία κλπ. κλπ. οι δορυφόροι μπορούν να δώσουν ένα σωρό χρήσιμες πληροφορίες. Στην τέως Γιουγκοσλαβία υπήρχε παράδοση με τον Μαγκιόν για παράδειγμα και άλλους δορυφόρους. Εσείς σκέφτεστε να δημιουργήσετε και έναν ε, διαστημικό σταθμό που κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της ζωής του. Η Κίνα για παράδειγμα σχεδιάζει κάτι τέτοιο. και τι σκέφτεστε για έναν σταθμό εκτόξευσης. Πολλοί ανταγωνιστές μας και εταίροι μας ανά τον κόσμο έχουν τέτοιους σταθμούς εκτόξευσης. Τέλος. Ποιο είναι το ποσοστό εξωτερικών πελατών της ESA. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλους ευρωβουλευτές, συναδέλφους. Η κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι προλαλήσαντες, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε με μεγάλη ενεργητικότητα. Βλέπω ότι υπάρχει πράγματι αυτή η δέσμευση από την πλευρά των Επιτρόπων και θέλω να του ευχαριστήσω. Μία δεύτερη παρατήρηση. Ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος είναι δύο σημαντικά εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Πρέπει όμως να βρούμε το σωστό τρόπο να έχουμε μια επικοινωνία προς τους πολίτες μας σε σχέση με τον, ε, τα ωφέλη αυτών των προγραμμάτων. Μπορεί να υπάρξουν πολλά σημαντικά ωφέλη και εφαρμογές που θα προκύψουν από τον Κοπένικο και θέσεις εργασίες και αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες μας να τα γνωρίσουν και για να μπορεί να υπάρξει πραγματικά υποστήριξη προς τα εγχείρηματα αυτά. Αυτό ισχύει λοιπόν και για τον Κοπέρνικο και για τον Γαλιλαίο. Πρέπει λοιπόν αυτά τα προγράμματα να γίνουν λειτουργικά για να φέρουν τους καρπούς που θέλουμε να αποδώσουν. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά ώστε να φτάσουν σε λειτουργικό στάδιο, αλλά κυρίως να κατανοήσουμε όλοι ποια είναι τα τεράστια οι τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών, ότι είναι προγράμματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ωφέλεια και θα δημιουργήσουν και θέσει εργασία στις νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, ψυχωμένη παρέμβασή σας υπέρ αυτών των πρωτοβουλειών. Είχαμε ακούσει και την προηγούμενη χρονιά τον ε, Επίτροπο Σέρτσοβιτς και την κυρία Μπιενκόφσκη, αλλά και τώρα χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δεσμευσή του. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Λιμπάτσκα. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση του θέματος αυτού, πολύ ενδιαφέρουσα η διαστημική στρατηγική. Έχω ερώτηση για την κυρία Μπιανκόφσκα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η διαστημική στρατηγική. Θέλουμε η διαστημική μας βιομηχανία να είναι καινοτόμος. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ε, ένα εργατικό δυναμικό με πάρα πολλά προσόντα ποιοτικά. Σε πολλά πανεπιστήμια, όπως και στη χώρα μου, ε, δημιουργούνται σχολές οι οποίες ε, θα προσφέρουν εκπαίδευση για αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Επίτροπε, αναφερθήκατε στη δήλωση που υπεγράφει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος για αυτή τη διακήρυξη, αυτή τη δήλωση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μνήμα εκεί για την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για νέους από όλα τα πανεπιστήμια, από όλη την Ευρώπη οι οποίοι θα εκπαιδεύονται στον τομέα αυτό, στη διαχείριση του διαστήματος και στην εκμετάλλευση του διαστήματος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι είναι επόμενος και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Εκτιμώ τις φιλοδοξίες μας για το διάστημα, κυρίως και σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές. Η διαστημική ε, στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την υποχρεωτική σχέση κόστος ωφέλους που αφορά όλα τα προγράμματα. Αυτό το κάναμε κατά το για το Γαλιλαίος. Ε, πολύ το κόστος του Γαλιλαίου κατά το παρελθόν. Πριν πάμε όμως στη, στο διάστημά μας, μείνουμε στον πλανήτη. Δράτω τις ευχές παρουσίας σας κύριε Επίτροπε, καταχρώμε μάλλον και τις παρουσίες σας, να θέσω ένα άλλο ερώτημα που δεν θα σας ευχαριστεί είναι το σχέδιο απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΟΠΑΛ, την Ευρωπαϊκή αυτή τη γερμανική υπηρεσία για, και να αυξηθεί η συμμετοχή της Gazprom στην ΟΠΑΛ. Είστε ελεύθερος να μην απαντήσετε, διότι είναι στο πρόγραμμα αυτό το θέμα, αλλά επίσης αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε ελεύθερα στην ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζανονάτο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Αντιπρόεδρο του κ. Σεύκοβιτς και την Επίτροπο την κυρία Μιανκόφσκα για την παρουσίαση και για τη στρατηγική που παρουσίασαν. Είναι μια, ένα όραμα που συμμεριζόμαστε, απαραίτητη στρατηγική και την αναμένουμε άλλωστε. Τα προγράμματα Γαλιλαίος Κοπέρνικος, έγνους είναι θεμελιώδου σημασία ούτως ώστε το ευρωπαϊκό σύστημα να είναι ένα σύνολο που περιέχει εργαλεία για τις πτήσεις και για άλλες χρήσεις, η θεμελιώδου σημασία. Και σίγουρα έτσι θα μπούμε στην πρώτη γραμμή του πλανήτη όσον αφορά τεχνολογία. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, Πρόεδρε. Και χρειάζεται τώρα που έχουμε τον Τραμπ να ακόμα παραπάνω να έχουμε αυτόνομα συστήματα. Το λέω εν είδη αστεϊσμού. Έχω δύο ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Σύντομα, η πρώτη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν διευκολύνουμε την πρόσβαση των προϊόντων της αριθμικής βιομηχανίας στις αναδιόμενες αγορές. Αναφερθήκατε σε αυτό, θα ήθελα ε, και κάποιες ε, λεπτομέρειες. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού με άλλες δυνάμεις διαστημικές. Πώς μπορούμε να είμαστε και εμείς στο ίδιο επίπεδο. Στα πλαίσια της διαστημικής, του διπλωματίας πώς τίθεται το θέμα της εποπτείας και της αφαίρεσης των αποβλήτων ε, του διαστήματος και το θέμα της ε, κυβερνασφάλειας. Πολύ σημαντικό. Είναι αρχική από το αρχικό στάδιο της κατακτήσεως του διαστήματος ε, συσσωρεύτηκαν πάρα πολλά απόβλητα και συντρίμια και είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ποιο πλαίσιο θα προωθήσουμε τη διαστημική διπλωματία πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕΣΑ και με τις εθνικές αρχές και με τις υπηρεσίες ε, ε, Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Πώς θα υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία των διαφόρων φορέων όσον αφορά το διάστημα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζολίνιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Έχει μεγάλη σημασία η Διατλαντική Συμμαχία και συνεργασία στα θέματα αυτά, αλλά βέβαια έχει μόλις λάβει μια μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια τάξη με τις Αμερικανικές εκλογές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα γνώσης και λειτουργίας στο διάστημα. Ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος είναι πράγματι σημαντικά και εμβληματικά σχέδια που μπορούν να αποτελέσουν ένα άξονα για την ανάπτυξη και άλλων προγραμμάτων. Να υπάρξει λοιπόν ένα στερέωμα από τέτοια σχέδια. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Πορτογαλία θέλει να προωθήσει μια νέα πρωτοβουλία που λέγεται η Ατλαντική Συμμαχία που περιλαμβάνει και τα νησιά της Μαδέρας και των Αζωρών ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο τομέα της ε, τεχνογνωσίας και ιδιαίτερα στον τομέα του διαστήματος. Πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία ενός ε, κέντρου συλλογής δεδομένου, δεδομένα από, το διάστημα, παρακολούθηση λοιπόν διαστη, ε, διαστημικών αποστολών και δορυφόρων, που να παρακολουθεί στην περιοχή του, ε, των Αζωρών, της ε, Μαδέρας, του Καμποβέρδε, της περιοχής της Βόρειας Βραζιλίας κτλ. Τα αντικείμενα που κινούνται στο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει λοιπόν και περαιτέρω δυνατότητα συνεργασίας, ενισχυμένης συνεργασίας με την Ισπανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, <coughs> με αφρικανικές χώρες και τη Βραζιλία, με την Αμερικανική Νάσα και την Βραζιλιανή Υπηρεσία Διαστήματος. Πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει ως μια μορφή ενισχυμένης συνεργασίας, σύνδεσης βορανότου, στην καινοτομία και στη μελέτη του διαστήματος και στους συναφείς τομείς. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ε, επιτρόπους να συμπεριλάβουν και αυτό το σημαντικό σχέδιο στη διαστημική του στρατηγική. Ο κύριος Κόξ. Ευχαριστώ δύο ερωτήματα θα ήθελα να θέσω προς την Επίτροπο Βιενκόφσκα. Θυμάστε την ακρόασή σας κύριε Επίτροπε όταν σας είχα θέσει ένα ερώτημα για το αν μπορούσατε να εντοπίσετε ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα το οποίο θέλετε να καταργήσετε για να μειώσετε το άχθος των επιχειρήσεων. Τα δύο χρόνια που είσαστε επίτροπος, δεν ξέρω αν έχετε βρει κάποιο τέτοιο νομοθέτημα, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι αυτό το νομοθέτημα. Ή αν όχι, θα μπορούσατε να βρείτε κάποιο τέτοιο νομοθέτημα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με τη διαστημική στρατηγική η τωρινή στρατηγική συμφωνία ασφάλειας των Νορβηγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στον Γαλιλαίο για την παροχή υπηρεσιών. Ξέρω ότι οι προσπάθειες για συμμετοχή της Νορβηγία στα θέματα αυτά έχουν μόλις επαναρχίσει, Μπορείτε θα μας δώσετε κάποια επίκαιρα στοιχεία για αυτές τις συνομιλίες και να μας εξηγήσετε αν έχουν προκύψει προβλήματα σχετικά. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσίασή σας, η παρουσίαση της διαστημικής στρατηγικής ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα έχουμε και κάποια προβλήματα που αφορούν την ενέργεια. Εξού και η ερώτησή μου. Η ερώτησή μου αφορά την ενεργειακή πολιτική. Κύριε Επίτροπε, εδώ και δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μια απόφαση. Απόφαση να δεχτεί τη θέση του, της γερμανικής ρευμαστικής αρχής όσον αφορά την πρόσβαση της Gazprom, τη μεγάλη συμμετοχή της Gazprom, να φτάνει στο 80%. Εάν δεν αγοράσει κανείς το υπόλοιπο 20%, η Gazprom θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για δικές της ανάγκες και να ενισχύσει έτσι τη θέση της όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η Gazprom δεν είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, είναι σαφές ότι είναι πολύ καλή απόφαση αυτή για την εταιρεία. Αυτή η κατάσταση λοιπόν και το ότι είναι παρόν εδώ επίτροπος με οδηγεί στην κάτω ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έρευνα όσον αφορά τις συνέπειες της απόφασης αυτής. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια απόφαση η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του φυσικού αερίου που παραδίδει Γκάσπρομ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τι συνέπειες έχει αυτό για την διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα σχέδια της Γκάσπρομ όσον αφορά την αύξηση ε, δυναμικού χωρητικότητας του Nord Stream ένα, επιβεβαιώνει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η απόφαση θα οδηγεί σε αύξηση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τρίτο, και πιο σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέταση τις επιδράσεις που έχει αυτή η απόφαση στην αγορά κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ και θα το εκτιμούσα αν ο κύριος Επίτροπος θα έχει την καλοσύνη να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις που αφορούν αυτά τα θέματα, γιατί είναι σημαντικές. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν ε, άλλες ερωτήσεις. Συνάδελφοι, ο κύριος Γκέρεκ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγγίξαμε κάποια θέματα γεωπολιτικής φύσεως. Θα παραμείνω λοιπόν και εγώ σε αυτό το τομέα. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Η υπηρεσία θα επικεντρωθεί κυρίως επί τεχνολογίας ε, πληροφορικής, τεχνολογιών πληροφορικής. Οπότε θα έχουμε μικρούς δορυφόρους και δεν θα έχουμε έναν μεγάλο σταθμό για να δούμε, να κάνουμε πειράματα πώς λειτουργεί η διαστημική τεχνολογία σε συνθήκες ελλείψεως βαρύτητας. Η, ε- η, η ΕΣΑ, η δική μας υπηρεσία, πώς θα συνεργαστεί με την αντίστοιχη ρωσική υπηρεσία που αναφέρθηκε που χειρίζεται το σταθμό, τη βάση. Θα ήθελα να σας πω ότι προκαιρού είχα εμπλακεί εγώ ο ίδιος στην κατεργασία νέων ε, κραμάτων και η συνεργασία μας τότε ήταν πολύ καρποφόρα. Υπάρχει νέος, ε, νέο πεδίο συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ο, Κρίστιον, ο κ. Κρίστιαν Έρλερ έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Σα φαίνεται παράξενο να το λέει αυτό ένα Γερμανός. Αλλά πιστεύω ότι το Nord Stream είναι ένα λάθο. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκπληκτικό το ότι υπάρχει μια τέτοια αντίσταση από τους συναδέλφους της Ανατολική Ευρώπης. Και αυτό το οποίο θέλουν ζητά να υπάρξει περισσότερη κοινή θέση για τα ενεργειακά θέματα. Εγώ νομίζω ότι το Nord Stream δημιουργεί μια, ένα πρόβλημα για την Ενεργειακή Ένωση, αλλά η Κομισιόν δεν έχει πει τίποτα για όλα αυτά, έχει αφήσει την έγκριση να γίνει από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή αυτή πολιτική, όπως πολύ σωστά το έχει ζητήσει αλλά φυσικά αυτή η πολιτική δεν υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα ήθελα λοιπόν ποιε είναι οι εκτιμήσεις της ε, Κομισιόν για το αν θεωρεί πράγματι το Nord Stream. Προβληματικό και αν εξάλλου έχει κάποια δικαιώματα να παρέμβει στη διαδικασία έγκρισης αυτού του αγωγού. Ευχαριστώ πολύ, Αγίου Πρόεδρος. Κύριε Αντιπρόεδρε, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορούμε να, με τη συνάδελφο να μοιραστούμε τις ερωτήσεις. Θα κάνω την πρώτη προσπάθεια και μετά θα απαντήσω για το θέμα Opal και Nord Stream. Το πρώτο ερώτημα του κυρίου Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που δώσατε όσον αφορά τις αισθημικές επιστήμες στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος εξεπλάγει τα μάλα όταν ήμουν στη Silicon Valley και προσεκλήθη στις εταιρείε εκεί με μικρές ή μεγαλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις. Είχαμε κοινή συνεδρίαση εκεί και πήγαμε την Λεσβίατα και ανακαλύψαμε ότι πάνω από, τις, από τους μισούς ανθρώπους που συναντήσαμε στις ΗΠΑ και εδώ στην Ευρώπη είναι Ευρωπαίοι. Εκπαιδεύονται στην Ευρώπη, μελετούν στα πανεπιστήμια μας, μελέτησαν στα πανεπιστήμια, ανέπτυξαν φανταστικά προγράμματα, αλλά μας λένε θα θέλαμε να μείνουμε στην Ευρώπη, το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Κεφάλαια κινδύνου, δυνατότητα επιμερισμού του κινδύνου και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε πραγματικά υπέροχα προϊόντα φοβερή υψηλή τεχνολογία και θα θέλαμε να το κάνουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχο μα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Θα με ρωτήσετε γιατί είμαστε δύο εδώ παρόντε. Εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται οριζόντια επικοινωνία. Γι' αυτό συνεργαστήκαμε στενά με τη Λισμπέτα, αλλά και με άλλου επιτρόπου. Θέλουμε και ο Γιώργη Κατάινε να μα βοηθήσει να δημιουργήσουμε αυτό το μέσο για την ε, χρηματοδότηση κινδύνου. Θα πρέπει και να συνεργαστούμε και με τον κύριο Έτιγκερ. Όταν φτάσουμε στα τηλέφωνα πέμπτη γενιά, 5G, να βρούμε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, τι χρειαζόμαστε από του δορυφόρου ε, πώ καλύπτουμε και τι απομακρυσμένε και αεροκατοικημένε περιοχέ. Θέλουμε να μιλήσουμε για με οδήγηση, συνδεδεμένα αυτοκίνητα, ε, με τους δορυφόρους, ε, τα ε, τρένα υψηλής ταχύτητας. Και εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η δορυφορική κάλυψη. Πρέπει να λάβουμε αυτά υπόψη. Μπορώ να αναφέρω πολλού συναδέλφους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συμμετάσχουν και ο Κάλλος Μόιδα. Αν μιλήσετε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, θα σα πούν ότι υποστηρίζουν τον ορίζοντα 2020 και άλλα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχουν πολλοί ερευνητικοί μας φορείς και αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα ήταν δύσκολη η ζωή των ερευνητών. Θα πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε για να προωθήσουμε σημαντικότατα προγράμματα στο μέλλον. Από αυτά που είδε ο Γιάννους είδαμε ότι ήταν πρώην επίτροπος ε, υπεύθυνο για οικονομικά και του αρέσει η ανάλυση κινδύνου και σχέση κόστο-οφέλου. Θέλαμε να σας δώσουμε καλά στοιχεία να σας αποδείξουμε ότι ο τρόπος ότι τα χρήματα που επενδύεται στα εθνικά προγράμματα επιστρέφουν 7 ευρώ στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι ποιοτική ανάπτυξη. Ε, είναι ε, τεχνο, ε, υψηλής τεχνολογίας αυτή η βιομηχανία, ποιοτικές της απασχόλησης και έτσι η Ευρώπη θα είναι σε ύψιστο επίπεδο όσον αφορά τι νέε τεχνολογίε που χρειάζεται και πρέπει να αναπτυχθούν. Συμφωνώ με τον κύριο Ρούμπικ, θα πρέπει να συζητούμε μεταξύ μα οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί σα και μαζί με άλλου σημαντικότατου φορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω την Utelsat, Εθνική Υπηρεσία Διαστήματο, ε, Εθνική Υπηρεσία Διαστήματο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και με την NASA. Ε, θα δείτε ότι έχουμε συνεργαστεί με διάφορους σε αυτό τον τομέα. Όλοι εκτιμούν το νέο πνεύμα συνεργασίας. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να παγιώσουμε και να προωθήσουμε στο μέλλον. Ο κ. Νίκ αναφέρθηκε στη σημασία του να προσγειωθούμε, αν θέλετε, ως όλα την προσέγγιση μας. Να δείξουμε στον κόσμο παραδείγματα συγκεκριμένα, απτά. Τι όφελος αποκομίζουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες από τα προγράμματα. Και ευχαριστώ και την κυρία Νόινχάουζεν που μας ρώτησε πώς να ξεκινήσουμε στους πολίτες τι ακριβώς πληρώνουν. Πρέπει μαζί, μαζί σας να κινηθούμε, να χρησιμοποιήσουμε σαν πρεσβευτέ τη διαστημική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, να κινηθούμε με του εθνικού φορεί. Θέλουμε στατική επικοινωνία, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ούτε ένα κινητό τηλέφωνο, ούτε μία, ένα τραπεζικό έμβασμα, ούτε ένα τρένο υψηλή ταχύτητα θα λειτουργούσε σήμερα στην Ευρώπη χωρί την δορυφορική τεχνολογία. Αν υπήρχε κάποια τεχνική δυσκολία ή κατέρε το σύστημα GPS, θα βλέπαμε πόσο εξαρτώμεθα από τι τεχνολογίε και γιατί οι Αμερικανοί ακόμα και προχθές δέχτηκαν ότι είναι καλό να υπάρχει συμπληρωματική δυνατότητα που θα παράσχει το Γαλιλαίος στην αγορά. Μεγαλύτερη ακρίβεια, πιο καινούργια τεχνολογία και πιο ποιοτικέ ε, υπηρεσίες. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και συγκεκριμένα παραδείγματα. Με συγκίνησε μια νεοφυής ισπανική εταιρεία που μας εξηγούσε ότι χάρη στη νέα ακρίβεια του Γαλιλαίου θα μπορούν να αναπτύξουν ειδικέ συσκευέ για να βοηθήσουν του ανθρώπου που έχουν πρόβλημα όραση. Που θα μπορούν τώρα να περπατήσουν χρησιμοποιώντα αυτέ τι συσκευέ και να περπατούν στην πόλη και στην ύπεθρο. Διότι το δορυφορικό σύστημα θα είναι τόσο ακριβέ που με αυτή τη συσκευή που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που δεν βλέπουν, θα μπορούν να περπατούν σχετικά ελεύθερα. Και αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που θα βοηθήσει πάρα πολλού ανθρώπου στην Ευρώπη, θα του δώσει μια νέα ελευθερία. Είναι συγκεκριμένο παράδειγμα και είμαι σίγουρο ότι θα το καταλάβουν, θα το στερνιστούν οι άνθρωποι. Και έχουμε λαμπρά νέα μυαλά στι νεοεφύσει ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και σύντομα πιστεύω θα έχουν πολλέ τέτοιε λαμπρέ ιδέε, παρόμοιε όπω αυτή που ανέφερα. Ο κ. Σανόφσκι αναφέρθηκε στο Brexit. Αν επιτρέπετε θα συνεχίσω αγγλιστή διότι αφορά αυτό που θα πω του Βρετανού φίλου μα. Όπω γνωρίζετε όλοι περιμένουμε να δούμε Ποιες θα είναι οι παράμετροι που θα θέσει η Βρετανίδα Πρωθυπουργό στους ε, Ευρωπαίους ομολόγους της για διαπραγμάτευση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιος είναι ο ρόλος του, της Βουλής του Κοινοτήτων, τι γίνεται με το Ανώτατο Δικαστήριο. Θα υπάρξουν και κάποιες νομικής φύσεως εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα πρέπει να είμαστε αρκετά υπομονετικοί. Να δούμε ε, ποια θα είναι η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί από, το, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για, το, για τα δύσκολα αυτά θέματα για όλους μας. Τι να σας πω τώρα για τον διαστημικό τομέα. Να σας πω το εξής. Όταν ήμουνα στο Συμβούλιο της ΕΖΑ, όπου εκπροσωπούνται όλες οι υπηρεσίες διαστήματος και συζητούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς συνεργαζόμαστε μαζί με τη Λεσβέθα για τη στρατηγική, Μία, ένα από τα θετικότερα, ε, θετικότερες υποστηρίξεις είχαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. να συμμετάσχουν στην συνεργασία, αναγνώρισαν ότι είναι ποιοτική προσπάθεια που καταβάλουμε ε, και είμαι σίγουρος ότι ανεξάρτητα το θέμα των συζητήσεων για τον Brexit, η, η Βρετανική Υπηρεσία Διαστήματος θέλει να συμμετάσχει, θα θέλει να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν πολύ από το γενικό τόνο και τις παραμέτρους των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Πολύ δύσκολο τώρα να κάνουμε εικασίες πώς θα πάνε τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε ε, καταρχάς ε, τη θέση της Βρετανικής κυβερνήσεως. Υπάρχει όμως καλή θέληση, αυτό ήθελα να πω από την πλευρά της αντίστοιχης Βρετανικής υπηρεσίας. Τώρα, αν αυτή η στρατηγική ε, είναι αρκετά ελκυστική, αυτό που έπρεπε να αποδείξουμε πιστεύω σε εσά και στο κοινό ήταν το εξής χειριζόμαστε μια υποδομή, προγράμματα προς καθημερινή χρήση των ε, πολιτών και θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο στεναροί εξηγώντα τη σημασία αυτών. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι άλλο. Ε, χωρίς να είμαστε τόσο σημαντικοί πελάτες, χωρίς να έχουμε τόση σημαντική στήριξη από πλευρά δημοσίων χρημάτων της ΕΣΑ, δεν θα μπορούσε η ΕΣΑ να προχωρήσει προς πιο ελκυστική εξερεύνηση του μακρινού διαστήματος, του βαθέως διαστήματος. Και ΕΣΑ σίγουρα θα παρουσιάσει σχετικό έγγραφο, περιμένει να δει ΕΣΑ πρώτη δική μας στρατηγική, ήθελε να υπογράψει την κοινή δήλωση μαζί μας, και χαιρόμαστε που εγγράφει, δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο. Θέλει να παρουσιάσει η υπηρεσία αυτή το έγγραφο για τη μελλοντική εξερεύνηση του ε, διαστήματος, του απόμακρου διαστήματος και θα το παρουσιάσει αργότερα του χρόνου. Ε, άρα θα παρουσιάσουν προγράμματα πιο ενδιαφέροντα, πιο ελκυστικά. Ε, και θα τύχουν σχολείων. Ο κ. Κόλιτσεκ έθεσε άλλο ερώτημα. Προστασία δεδομένων, συλλογή δεδομένων. Και πόσες επιχειρήσεις απ' έξω από την Ευρώπη ε, εμπλέκονται στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. Δεν έχω στοιχεία ακριβή. Όσον αφορά τον εμπορικό διαστημικό τομέα, όπω τα αποκαλούσα, σχεδόν ο ίμιση τομέα καλύπτεται από την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. Βλέπετε πόσο ισχυροί είμαστε στα θέματα αυτά. Όσον αφορά τον πολιτικό διαστημικό τομέα, είμαστε νούμερο ένα στον κόσμο, θα έλεγα. Διότι στι ΗΠΑ, στην Κίνα και την Ινδία ο διαστημικός χώρος καλύπτεται σε το βαθμό από το στρατιωτικό τομέα. Και εδώ έχουμε ε, πολύ ισχυρή κάλυψη πλευράς ε, του πολιτικού τομέα, όχι του στρατιωτικού. Τώρα, αν με επιτρέπετε τώρα να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα λοιπόν ε, στο τέλος, στα τελευταία μου λεπτά, να αναφερθώ στο ΟΠΑΛ και στο Nord Stream τις ερωτήσεις σχετικέ. Είμαι στην Επιτροπή Ήτρε, ξέρω ότι παρακολουθείτε αυτά τα θέματα με μεγάλη προσοχή και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω επ' αυτών, παρόλο που συζητούμε ένα διαφορετικό θέμα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το OPAL, αυτό ήταν πολύ ευαίσθητο και δύσκολο σαν απόφαση που έπρεπε να ληφθεί, διότι πρέπει να σεβαστούμε και τους δικούς μας κανόνες. Έπρεπε επίσης να εξετάσουμε και το όλο ιστορικό όταν κατασκευάστηκε το Nord Stream 1 μετά τη μεγάλη κρίση του φυσικού αερίου του 2009, τότε ήταν κοινοφελές έργο το Nord Stream 1 και ήταν ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο ενεργειακό πακέτο και λόγω αυτών των αιτίων υπήρχε μια εξαίρεση που δόθηκε στον πετρελαγωγό, τον αγωγό μάλλον Όπαλ που αποτελεί από δύο τμήματα. Ένας αγωγός πάει από τη θάλασσα Προ έναν κόμβο κοντά στο Βερολίνο για το φυσικό αέριο και από αυτό το κόμβο του φυσικού αερίου πάει στα τσεχικά σύνορα. Και τι νομίζω που είναι κοινό σφάλμα είναι ότι πιστεύουμε ότι η Gazprom έχει 50% νομίζω όριο ε, τη χρήση του αγωγού. Δεν αληθεύει. Η Gazprom είχε 100% τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον αγωγό όπαλ υπό έναν όρο την Gazprom θα επέλεγε πρόγραμμα δημοπράτησης του φυσικού αερίου τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο, λιγότερο από το 10% της χωρητικότητας ε, του εν λόγω ε, αγωγού φυσικού αερίου. Μετά από αρκετά χρόνια ε, η Bundesnetz Agentur, ο γερμανικός μυστικός φορέας, πρώτη αλλαγή τη εξαίρεση. Οπότε εμεί είχαμε τρει επιλογές. Πρώτη επιλογή, να μην δράσουμε. Εν τη αυτή περιπτώσει η πρόταση τη γερμανική θα ήταν να ανοίξουμε το αγωγό κατά 5% σε τρίτες, τρίτους φορείς τον πρώτο χρόνο και 4% το δεύτερο ε, χρόνο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει δεκτομία. Δεύτερη επιλογή, η οποία προετάθη να έχουμε απορρίψει την πρόταση αυτή του ΟΠΑΛ. Τότε όμως και το αναλύσαμε πολύ προσεκτικά. Δεν είχαμε μία πραγματική βάση για να μπορέσουμε να το απορρίψουμε, γιατί θα ήταν απόρριψη μόνο για πολιτικούς λόγους και σε οποιοδήποτε δικαστήριο θα χάναμε μία προσφυγή και θα ήμασταν και θα μας φέρουν και ενώπιον του πάνελ του <clears throat> ΠΟΕ και όπου ήδη μας έχουν, έχουν κάνει προσφυγή εναντίον μας γιατί μας κατηγορούν ότι εφαρμόζουμε την ενεργειακή <clears throat> ε, ένωση με πολιτικά κριτήρια. Η Bundesnetzagentur λοιπόν ε, έδωσε μια πρόταση η οποία είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα, πολλές σελίδες, πολύ δυσανάγνωστου κειμένου γιατί είναι... Αν πρέπει όμως να απλοποιήσω λιγάκι τα πράγματα αυτά, όλα αυτά σημαίνουν ότι 50% του αγωγού αυτού είναι για την Gazprom και το άλλο 50% αυτό που θα φέρνει λοιπόν από τον κόμβο κοντά στο Βερολίνο προς την Τσεχία θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε τρίτους φορείς αλλά πολύ περισσότερο από ό,τι στο αρχή. Κατά 20% γενικά. Επομένως, επιτυχάνουμε να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο καθεστώς από ό,τι είχε προταθεί αρχικά και για πρώτη φορά <clears throat> ανοίγουμε αυτό τον αγωγό σε τρίτους φορείς που δεν είναι κατά ανάγκη η Gazprom και να μπορούν να μεταφέρουν λοιπόν από το Βερολίνο προς την Τσεχία. Κάναμε λοιπόν ό,τι, ό,τι μπορούσαμε περισσότερο. Υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης που σημαίνει ότι αν δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για περισσότερη μεταφορά φυσικού αερίου θα είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την τεχνική εφικτότητα της χρήσης του αγωγού για αυτό το στόχο, γιατί τότε θα χρειάζονται και περαιτέρω σταθμοί συμπίεσης και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αυτήν την δυνατότητα. Μα τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα για την Ουκρανία ή για τη διέλευση του αγωγού μέσω της Πολωνίας. Το ελέγξαμε και αυτό και είναι γεγονός ότι σε ό,τι μπορούμε να διακριβώσουμε τα συμβόλαια διέλευσης για την Ουκρανία και άλλες χώρες θα πρέπει να είναι ε, συμβόλαια μακροχρόνια με συγκεκριμένα σημεία παράδοσης. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι θα προκύψει μια απότομη μείωση στους όγκους φυσικού αερίου που πηγαίνουν προς την Ουκρανία ή μέσω και ξέρετε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ μιλάω μονάχα εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχω μια ομόφωνη υποστήριξη σε αυτό από όλα τα κατημέλια από του Υπουργού Οικονομικών, Εξωτερικών, ότι η διατήρηση των δρόμων διέλευση μέσω της Ουκρανίας μετά και το 2020 είναι μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε πει και στη ρωσική πλευρά. Είναι μια προσέγγιση που υποστηρίστηκε από τη Γερμανία. Και αυτό αναφέρεται κάθε φορά που συζητούμε το θέμα αυτό. Εάν λοιπόν πρόκειται να υπάρχει περισσότερος όγκος φυσικού αερίου, ο οποίος θα ερχόταν σε αυτόν τον κόμβο κοντά στο Βερολίνο, θα ήταν ε, σταδιακά δυνατό. Βέβαια υπάρχουν διάφορε εκτιμήσει για το πόσο μπορεί να είναι αυτός ο πρόσθετο όγκο λόγω της ικανότητας μεταφοράς του αγωγού για τη δυνατότητα χρήσεώς του. Αποφασίσαμε λοιπόν να έχουμε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο επιπλέον. Θεωρούσαμε ότι αυτό όμως αυτή η ποσότητα θα πίνει περισσότερο στην δυτική αγορά παρά στην αγορά της κεντροανατολικής Ευρώπης. Και σε ό,τι αφορά το Nord Stream, διαπίστωσα πέρσι ότι είναι απαραίτητο να είμαστε πολύ προσεκτικοί για οποιοδήποτε από αυτά τα Nord Stream, το νότιο, το βόρειο, το ανατολικό, το δυτικό, γιατί πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν, πότε αλλάζουν τα consortium. Και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντικό βέβαια για την Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε στην πεποίθησή μας ότι η ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα από την διαφοροποίηση. Είναι καλύτερα λοιπόν να είναι όλοι ανοιχτοί σε διασυνδέσεις με οποιοδήποτε πάροχο ενέργεια στην Ευρώπη και οποιοδήποτε παρέχει ενέργεια στην Ευρώπη θα πρέπει να σέβεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό αφορά και το Nord Stream και οποιασδήποτε τέτοιες διασυνδέσεις θα πρέπει να ισχύουν και αυτό θα πρέπει να αφορά και το υπεράκτητο τμήμα του αγωγού Nord Stream. Αν λοιπόν λειτουργήσει αυτό το σύστημα και το σχέδιο, ποιε είναι οι παράμετροι, θα πρέπει να το δούμε αυτό, να το συζητήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συγγνώμη, αλλά θέλω να απαντήσω απλώ και αυτό το δεύτερο σύνολο ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι για όλα, ακόμα και για μακρύς ομιλίε. Η κυρία Επίτροπος τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο ήταν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ θα είμαι κάπως πιο σύντομη, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Η στρατηγική είναι μια συνολική δουλειά από διάφορα σώματα, όργανα και πολλούς εταίρους. Και αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί και η εταίροι βρήκανε καλή τη στρατηγική αλλά και όλη τη διαδικασία προετοιμασίας της. Αυτή η προετοιμασία ήταν χρήσιμη. Χρησιμοποίησαμε την γνώση και η βιομηχανία εκτίμησε όλος ιδιαίτερος τη διαδικασία αυτή. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στη στρατηγική. Ο Μάριος είπε, και είναι ένα απλό παράδειγμα, ότι ένα ευρώ για το διάστημα δεν είναι πίσω 7. Ίσως και περισσότερα αν βάλουμε υπόψη μας ε, το ΕΠ, την απασχόληση. Επίσης, το άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να υποθεί. Γιατί είχαμε αυτή την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εμπορική αγορά όσον αφορά τα δεδομένα του διαστήματος και για τη βιομηχανία βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι υπεύθυνη για την ε, ανακάλυψη του διαστήματος και την εκμετάλλευση του διαστήματος. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ρωτήσατε ποια θα είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλουμε να φτιάξουμε μία λυσίδα αξιών όσον αφορά το διάστημα και για τις εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο διάστημα, τις καινούργιες, τις startups, με νέες πλατφόρμες διάδοσης των δεδομένων. Να μην πρέπει να κατεβάζουν όλα τα δεδομένα, αλλά να μπορεί να υπάρχει ένα software που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε διάφορα clouds και σε διάφορους ε, servers ώστε η καινοτομία να καταστεί πιο εύκολη. Είμαστε εδώ λοιπόν για την εμπορική χρήση των δεδομένων και για τη δημιουργία της αγοράς για τις startups και για τη δημιουργία της αγοράς για τις εφαρμογές του διαστήματος. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί δουλεύουμε εδώ και καιρό δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελκυστική ή όχι αυτή η στρατηγική. Συμφωνώ συμφωνω όμω για το ότι δεν υπάρχει συνδυτοποίηση στην κοινωνία για το πόσο σημαντικό είναι το διάστημα. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου και συνέντευξη με τον Μάρος και λέγαμε πόσο πολύ μας ενθουσιάζει αυτή η υπόθεση του διαστήματος, γιατί εμείς εδώ και καιρό δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιο είδου στρατηγική επικοινωνίας γιατί εμείς σε αυτή την αίθουσα ξέρουμε πώς χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας ε, τις εφαρμογές του διαστήματος. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία, μόνο που δεν το ξέρουν. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Και πρέπει να το πούμε με πιο δυνατή φωνή από εδώ και πέρα. Επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί επανέρχομαι σε αυτό το κομμάτι το εμπορικό και το οικονομικό, πρέπει στην ε, ανακοίνωση της στρατηγικής μας να απευθυνθούμε στις επιχειρήσεις, στις ε, μικρομεσαίες, στις startups και θέλουμε τη δικιά σας στήριξη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ε, συνεντεύξεις και διασκέψεις και είχαμε πολύ ενθουσιώδη ανταπόκριση. 12 εκατομμύρια έχουμε δαπανίσει και πρέπει να αιτιολογήσουμε, να δικαιολογήσουμε ήταν και είναι χρήματα τα οποία δαπανώνται καλά. Με ρωτήσατε επίσης για τους σταθμούς, τους σταθμούς. Ο κύριος Κοχλίκτσετ ρώτησε Λοιπόν, όχι. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκεφτόμαστε να φτιάξουμε έναν διαστημικό σταθμό η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία θα μπορούσε να το κάνει. Επαναλαμβάνω ότι εμείς ασχολούμαστε με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά στην ε, πραγματικότητα την οικονομική. Τα προσόντα, οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να προωθήσουμε την ιδέα αυτή της κατάρτισης για νέους, για φοιτητέ. και σίγουρα θα το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το μέλλον. Για το SST, στα πλαίσια και των Αμερικανικών εκλογών δραστηριοποιούμεθα στη συζήτηση όσον αφορά τα διαστημικά απόβλητα. Πολλά εξαρτώνται και εδώ από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πέντε χώρες μέλη με τις οποίες συζητάμε που θέλουν να επεκταθούν γεωγραφικά. Μετά θα δούμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με ένα σύστημα συνειδητοποίησης ώστε να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις ε, επιθέσεις, ε, το γενικότερο κλίμα και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα διαστημικά απόβλητα. Κύριε Λεβαντόσκη, το έγραψα ότι ναι, θα χρησιμοποιήσουμε το γαλαξία προς όφελος της οικονομίας μας. Ναι, δεν ήταν ερώτηση για το διάστημα. Για την ερώτηση του κύριου Φόξ. Στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο έχουμε κάνει πολλά θετικά για να μην παράξουμε νέο κανονισμό. Για παράδειγμα για τη συνεργατική οικονομία. Βλέπετε είμαστε τέρι αλλά βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μα ζητήθηκε να προχωρήσουμε όσον αφορά την συνεργατική αυτή οικονομία. Όμως υπάρχει πάρα πολλή νομοθεσία γι' αυτό και εμείς αυτό ακριβώ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τόσο πολλές ρυθμίσεις που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά που υπάρχουν υπέρ τη συνεργατικής οικονομίας και να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Έχουμε και μια νέα ε, προσέγγιση όσον αφορά την ε, επιβολή, τη συμμόρφωση, την ευφύ συμμόρφωση. Όσον αφορά τον κανονισμό, δουλεύουμε σε δύο τομείς copyright, πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή, και ίσως μπορέσουμε να μειώσουμε κάποιους κανονισμούς εκεί, και REACH, που είναι, ξέρετε, τα χημικά στην αεροπλοεία. Για τη συνεργασία μας τώρα με τους εταίρους μας, ελπίζω δεν θα αλλάξει τίποτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Ρωσία ο τελευταίος διάλογος που είχαμε ήταν τον Ιούνιο του 2013. Έκτοτε δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις για το πότε θα έχουμε την επόμενη συνάντηση. Βέβαια, συνεργαζόμαστε, αλλά μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος για το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και... Σας ευχαριστώ και τους δύο, αμφότερους και τους δύο. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι στις 28 και 29 Νοεμβρίου και σε αυτήν θα προσκαλέσουμε την ΕΣΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, για φυσικά και τον αντιπρόεδρο κύριο Σεύτσοβιτς και την κυρία Μπιενκόφσκη και θα συζητήσουμε το θέμα της εφαρμογής της στρατηγικής μας το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εκκίνηση της στρατηγικής για το διάστημα που είναι πάρα πολύ σημαντική και συναρπαστική πρόταση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Thanks. Thanks a lot. And don't, don't, don't leave you this. with this leash to the NATO, to the NATO meeting. No. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τα παρόντα μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ, πρώην μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ,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 Ε, Φίλοι, αγαπητοί. Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Ο, για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και για την ανταλλαγή απόψεων είναι μια ε, συνάντηση τακτική, όχι αυτή που δεν είναι η πρώτη φυσικά τέτοια συνεδρίαση των ρυθμιστών στον τομέα της ενέργειας με τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε μονάχα τον διευθυντή της Acer και το πρώτο του Συμβουλίου των Ρυθμιστών αλλά και την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα αυτού και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και πρώην μέλος της Επιτροπής μας. Α, η κυρία Γιώργα Σίζελ. Έτσι δεν είναι Ρωμάνα. Καλά τα λέω. Ρωμάνα Γιώργα Σίζελη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε. Και αν θα ήθελες θα μπορούσες να ξεκινήσεις τη συζήτηση με τα δικά σου σχόλια, Γιορδάνα. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Ευχαριστώ, Γέρζη. Αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κάποιοι από εσά είναι και πρώην συνάδελφοί μου. Χαίρομαι που είμαι εδώ ξανά μετά από καιρό υπό διαφορετική ιδιότητα. Είμαι πρόεδρος του, του Διοικητικού Συμβουλίου της Acer. Να επενθυμίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μέλες. Πέντε διορίζονται από το Συμβούλιο, δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δύο από το Ευρωκοινοβούλιο. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη που διορίστηκα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο δεύτερος που διορίσατε είναι ο Τάμις, και έχουμε και δύο αναπληρωματικά μέλη που διώσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθηγητή Ούρε Λέπριχ και Αντόρι χόρχεβ Βιέργα Τεβασκονσέλο. Στόχος είναι να κατατίζουμε τον προπολογισμό, να ελέγχουμε την εκτέλεση αυτού, να θεσπίσουμε εσωτερικού κανόνες, να θεσπίζουμε ε, κανονισμούς, να διορίζουμε διευθυντή, επίσημα να διορίζουμε μέλη του του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενστάσεις και του Διοικητικού Συμβουλίου των Εθνικών Φορέων και να εκτελούμε την αποστολή μας ε, που ανατίθεται. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την έκθεση για την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό κάθομαι εδώ σήμερα. Να σας διαβιβάσω ένα μήνυμα. Αν μου δώσετε άλλο ένα λεπτάκι. Από όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, Ιανουάριο φέτος. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε σημαντικό θέμα. Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων. Σας διαβάζω το μήνυμα. Αυτό δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο τεχνικό πρόβλημα, αλλά πολιτικό πρόβλημα επίσης. Γιατί? Διότι η Ενεργειακή Ένωση είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες αυτής της θητείας. Το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια και η εσωτερική αγορά αυτών είναι βασικός πυλώνας της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτή η αγορά θα πρέπει να απελευθερωθεί και να ρυθμίζεται σωστά και να ελέγχεται σωστά και αποτελεσματικά. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι επικρατεί ακαιρεότης και διαφάνεια. Το θέμα των ανθρωπίνων πόρων είναι ζήτημα πολιτικό. Θα σταματήσω. Δεν μου αρέσει να καταχρώμε του χρόνου σας. Λάβετε το υπόψη σας όμως όταν θα ξανασυζητήσετε θέματα προπολογισμού την επόμενη φορά όταν θα συζητήσετε τη θέσπιση νέων κανόνων και την έγκριση νέων νομοθετημάτων. Προσβλέπω πράγματι σε συζήτηση των προβλημάτων μαζί σας και σε κάποια άλλη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Ευχαριστώ τα μάλα λέει και ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου. Ρωμάνα, έχεις περάσει 10 χρόνια στην Επιτροπή Ήτρε 2004-2014 Περνάμε λοιπόν στις επόμενες παρεμβάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλμπέρτο Ποτότσνικ, ο οποίος είναι διευθυντής της Acer. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά για μας να έχουμε και φέτος αυτή την ευκαιρία. Γίνεται έθιμο πλέον αυτό <clears throat> να παρουσιάσουμε τα στοιχεία της εκθέσεως μας παρακολούθησης. Η εκθέση αυτή δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί και εδώ είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε μονάχα μια σύντομη σύνοψη των πορισμάτων αυτής της ανάλυσής μας και των συστάσεων μας. Είναι η πέμπτη ετήσια έκθεση που δημοσιεύουμε και κοιτάζει λεπτομεριακά η έκθεση αυτή την πρόοδο για την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθών να <clears throat> εντοπίσει φραγμούς και εμπόδια στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και προτάσει για το πώς θα ξεπεραστούν αυτοί οι φραγμοί. Μερικά καλά νέα. Για πρώτη φορά μετά από το 2010, οι περισσότεροι καταναλωτές στην Ευρώπη <clears throat> εποφελούνται και εποφελήθηκαν ήδη πέρσι από χαμηλότερες τιμές. Αυτό δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της φιλελευθεροποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, διεθνείς τάσεις στην τιμή της ενέργειας, αλλά βλέπουμε οι περισσότεροι καταναλωτές να επωφελούνται. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα με τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Ισχύει επίσης για την κατανάλωση ηλεκτρισμού από βιομηχανικούς πελάτες. <clears throat> Αλλά δυστυχώς για τα νοικοκυριά Μόνο στα μισά Τιμέλη υπάρχει βελτίωση των τιμών ηλεκτρισμού, ενώ στα άλλα έχει αυξηθεί. Αλλά όπως βλέπετε από αυτό το γράφημα, οι τιμές καταναλωτών δείχνουν αυτή την τάση που αναφέραμε για πολλά χρόνια. Αλλά μας ανησυχεί ακόμα η σύνθεση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτή. Μειώνεται το τίμημα τη ενέργεια μέσα σε αυτού του λογαριασμού. Το κομμάτι λοιπόν αυτό το οποίο είναι το αδιαμφισβήτητο κομμάτι της, ε, του τιμολογίου που δεν μπορεί <clears throat> να τροποποιηθεί από τον ανταγωνισμό είναι πολύ σημαντικό και αν δείτε τώρα τον ηλεκτρισμό και δεν βλέπουμε εδώ πέρα τα νοικοκυριά ο ανταγωνισμός μπορεί να <clears throat> αναπτυχθεί μόνο για το 1 τρίτο του τιμήματος του ηλεκτρισμού. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εμποδίζεται ο ανταγωνισμός. Τα υπόλοιπα είναι τέλη για το δίκτυο και τέλη για την υποστήριξη των ανανεωσίμων ενεργειών που έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε ό,τι αφορά το μερίδιο της <clears throat> για το τίμημα της ενέργειας. Η δική μας λοιπόν σύσταση προς τα κάτι μέλη να το δουν το θέμα αυτό και να δουν σε ποιο βαθμό αυτές οι, αυτά τα τέλη για την υποστήριξη ανανεώσιμων ενεργειών και άλλων μηχανισμών θα μπορούσε να καλυφθεί με άλλους τρόπους και όχι μέσω πρόσθετων τελών για το τίμημα ενέργειας. Γιατί όπως είπαμε προηγούμενος αυτό ουσιαστικά εμποδίζει τον ανταγωνισμό. Αλλά βλέπουμε, όπως είπα προηγουμένως, και κάποια ωφέλη τα οποία φτάνουν σιγά σιγά στους <clears throat> καταναλωτές λόγω της ολοκλήρωσης της αγοράς χονδρικής στην ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα στην αγορά. Για το φυσικό αέριο λειτουργεί πολύ καλά <clears throat> αυτή η αγορά. Ίσως θυμόσαστε από πέρσι την κατάσταση που σας παρουσίασα που δεν ήταν τόσο θετική. Αυτή η διαφάνεια δείχνει το μέσο κόστος <clears throat> σε κάθε χώρα σε σχέση με τον ε, κόμβο των της υπήρου μας που είναι η Ολλανδική TTF. Οι χώρες που είναι κίτρινες είναι εκεί που υπάρχει ελάχιστη διαφορά, λιγότερο από ένα ευρώ. Το γαλάζιο εκεί όπου η διαφορά είναι μεταξύ ενός και τριών ευρώ και οι, οι σκούρες μπλε εκεί που είναι μεγαλύτερη κατά 3 ευρώ ή παραπάνω διαφορά. Γίνεται όλο και πιο κίτρινη η Ευρώπη. Πέρσι δεν ήταν κίτρινη η, Ισπανία, η Ελλάδα ήταν σκούρο μπλε και τώρα μόνο έχει γίνει γαλάζια. Λοιπόν, μπορούμε από αυτό το γράφημα να δούμε, από αυτό το χάρτη να δείτε ότι προωθείται, προχωρεί η ολοκλήρωση της αγοράς και αυτό το οποίο δεν έχει σημασία δεν είναι η απόσταση από την πηγή του φυσικού αερίου, αλλιώ θα ήταν κίτρινο το κομμάτι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά το πιο είναι, είναι πιο κοντά στις αγορές. Γι' αυτό έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να έχουμε κόμβους για το φυσικό αέριο, ώστε να είναι κοντά στις αγορές. Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά για το υπόδειγμα που ακολουθούμε, λειτουργεί πολύ καλά. Απλώς πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Στην περίπτωση του ηλεκτρισμού τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει σωστή κατανομή της ε, ικανότητος, <clears throat> της παραγωγικής ικανότητος. Βλέπουμε ότι κατά 84% χρησιμοποιείται ο παραγόμενος ηλεκτρισμός, αλλά <clears throat> μεταξύ ημερών και σε ό,τι αφορά την εξισορρόπηση έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Μα ενδιαφέρει λοιπόν να μπορούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια από εκεί που είναι φθηνότερη στα μέρη που έχει τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Υπάρχουν όμω διάφορα παράπονα που έχουν διατυπωθεί για τι χαμηλέ τιμέ των αγορών. Και εδώ βλέπουμε ότι. ότι έχουμε ένα πρόβλημα υπερβολικής ικανότητας σε πολλές αγορές. Βλέπουμε στην ε, Γερμανία και τις κάτω χώρες, βλέπουμε να εξαφανίζονται οι απότομες κορυφές στην, ε, αίτηση, στην ζήτηση ε, ενέργειας, βλέπουμε κυρίως χαμηλές τιμές. Αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί έχουμε υψηλή ικανότητα παραγωγής, χαμηλές τιμές στην αγορά ε, ενέργειας. Έχουμε λοιπόν ένα <clears throat> πρόβλημα χρημάτων τα οποία έχουν εξαφανιστεί και αυτό οδηγεί σε έλλειψη επενδύσεων και οι μηχανισμοί για την υποστήριξη της παραγωγικής ικανότητας το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι αυτοί μηχανισμοί δεν βασίζονται στη λειτουργία της αγοράς. Μεταφέρουμε λοιπόν πράγματα που έπρεπε να είναι στην ε, αγορά εκτός αγοράς και ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπα προηγουμένως ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ε, τιμής ενέργειας καθορίζεται στην αγορά και το περισσότερο είναι από <clears throat> τέλη. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι το να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς που δεν είναι μηχανισμοί της αγοράς θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, ιδίω αν αυτοί οι μηχανισμοί είναι εθνικού χαρακτήρα. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει είναι πόσο μεγάλο κομμάτι της υπάρχουσας ικανότητας χρησιμοποιείται σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρώπη. Ποιο είναι κομμάτι λοιπόν αυτής της ικανότητας το οποίο μπορεί να τύχει εμπορίας. Με την τωρινή διασύνδεση κατά μέσο όρο μόνο η 28% είναι αυτό το οποίο την χάνει εμπορίου. Εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το 100%, δεν είμαστε τόσο αφέλης, το μόνο το 28% είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Και ο φορέας μας προσπαθεί να δει <clears throat> πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπολογισμοί ικανότητος για να χρησιμοποιούμε ένα μεγαλύτερο τμήμα αυτής της ικανότητας για εμπορία. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σύντομη σύνοψη για το πώς λειτουργεί η αγορά, η χοντρική αγορά φυσικού αερίου λειτουργεί πολύ καλά. Στον ηλεκτρισμό έχουμε κάνει κάποιες προκλήσεις. Το επίπεδο λιανο, λιανικής αγοράς τώρα. Βλέπουμε ότι οι ρυθμιζόμενε τιμέ παραμένουν σε πολλά κράτη-μέλη. Και για τα νοικοκυριά, αλλά και πολλέ φορές και για την ίδια τη βιομηχανία. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμιζόμενε τιμέ εμποδίζουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Και πράγματι από πέρσι ο φορέας μας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ανταγωνισμού στις τιμές καταναλωτή, στις διαρκές τιμές, συγκρίνουμε τις τιμές σε διάφορες χώρες, είναι ένα σύνθετος και δεν θέλω να σας καταδαπανίσω το χρόνο σας με τις λεπτομέρειες. Πρόκειται για νέα διαφορετικές διαστάσεις. Όταν όμως συγκρίνουμε την επίδοση της λιανικής στην Ευρώπη και κοιτάξουμε πώς οι αγορές με απελευθερωμένες τιμές συνεχίζουν να ρυθμίζονται και αυτές που είναι σε μεταβατική περίοδο, βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός πάει πολύ καλύτερα όταν, έχουμε όταν δεν έχουμε ρυθμισμένες τιμές. Βλέπουμε επίσης τις ε, αλλαγές στις τιμές όταν ε, οι καταναλωτές μπορούν να αποφεληθούν από την επιλογή. Έτσι μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση και υπάρχει θετικός συσχετισμός και με άλλα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους οι καταναλωτές όταν αποφασίσουν αν θα αλλάξουν ή όχι προμηθευτή. Το καλό νέο είναι ότι όπως οριμάζει το θέμα, δηλαδή χώρες που έχουν απελευθερώσει νωρίτερα τον τομέα, η διαφοροποίηση στην προσφορά ενισχύεται. Έχουμε πιο πολλές προσφορές με πράσινο, πράσινη συνιστόσα, ανάλογα με το χρόνο της κατανάλωσης κτλ. Όλα αυτά βέβαια παίρνουν χρόνο. Αλλά για τις αγορές ήδη συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις. Οπότε αυτό που θέλουμε εδώ είναι οι χώρες μέλη να προωθήσουν την αποδοτική χρήση της ενέργειας στις υποδομές, εκμεταλλευόμενοι ακόμα περισσότερο την δυνατότητα εισαγωγής ε, δυναμικών τιμών. Δύο τελευταία σημεία τώρα για τις αλλαγές και για τις προσφυγές. Πρόκειται για την προστασία των καταναλωτών. Φυσικά και θέλουμε να προωθήσουμε την επιλογή για τον καταναλωτή, αλλά οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αλλάξουν και άρα να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες στις χώρες μέλη. Εδώ συνοψίζουμε τις νομικές διατάξεις και την πρακτική στις χώρες μέλη. Κατά μέσο όρο βλέπετε ότι οι χώρες μέλη συμμορφώνονται σε τρεις εβδομάδες. Φυσικά υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Και τελικά όταν πρόκειται για προσφύγες, οι περισσότερες έχουν να κάνουν με συμβατικά ζητήματα και ζητήματα τιμών. Εμείς ζητούμε να χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί μηχανισμοί διευθέτησης διαφορών. Όταν η αρχή, η αρμόδια δεν είναι εθνική, αλλά η εθνική έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, μπορεί να επιθεωρήσει την κατάσταση. Αυτά είχα λοιπόν να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και μια τελευταία παρατήρηση. Την έκθεση αυτή την ετοιμάζουμε εδώ και πέντε χρόνια. Κάθε χρόνο δηλαδή την κάνουμε. Του χρόνου θέλουμε να μικρύνουμε την έκθεση αυτή. Οι πόροι πρέπει να πάνε στον έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενική Διευθύντα. Έχουμε το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ρυθμιστών, τον Πρόεδρο του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου. Οπότε δεν ξέρω εσείς, the Mog, Πρόεδρος, θέλετε το λόγο. Ίσως ναι, καλό θα ήταν να μπορείτε να πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα είναι καλό που με προσκαλείτε. Σας ευχαριστώ και με τιμά το γεγονός ότι μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε τη θέση μας, αλλά θέλω να σχολιάσω λίγο σε αυτά που είπε ο συνάδελφος. Το έγγραφο αυτό 11 λεπτά βέβαια χρειάστηκαν για να δείτε τη διαφάνει, τις διαφάνειες, αλλά η δουλειά που έχει γίνει από πίσω από αυτές τις διαφάνειες καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερη. Αδική δηλαδή τη δουλειά που έχει γίνει αυτό το σύνολο διαφανειών. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς, η κατάσταση αλλάζει. Νομίζω λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε μια πραγματική αντίληψη του τι συμβαίνει στην αγορά. Δεύτερον, η παρουσίαση δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος στις τιμές, στην ε, δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή. Σίγουρα θα μπορούσε η κατάσταση να είναι ακόμα καλύτερη, αλλά είναι καλύτερη έτσι κι αλλιώ. Και αυτό θέλαμε να τονίσουμε. Και τρίτον, όσον αφορά τη συνεργασία, έχουμε τι δύο οργανώσει. Δεν ξέρω αν θέλω να είμαι πρόεδρο, δεδομένων των σημερινών αποτελεσμάτων. Πάντω, οι δύο οργανώσει συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Η ένταση που υπάρχει έχει να κάνει με το χρόνο τον οποίο μπορεί να διαθέσει κάθε εθνική ρυθμιστική ε, αρχή για να συνεισφέρει στο Acer. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε και εθνικές αρμοδιότητες. Οι πόροι είναι περιορισμένοι, οπότε θα βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Και ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι, ότι η λιτότητα έχει επισέρθει και σε μας. Και η πραγματικότητα το θέμα της ενέργειας είναι ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την αγορά και να επιβάλλουμε τις αποφάσεις. Η Επιτροπή σας μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Και η ομάδα επαφής. Έχουμε υποφεληθεί πραγματικά από τις προσπάθειες και από τα ψηφίσματα, από τις προτάσεις για τα δημοσιονομικά. Έχουν γίνει κάποιες μικρές βελτιώσεις, αλλά Κάθε φορά επιστρέφουμε στην πηγή. Και τέλος, κάποια στιγμή θα αποδειχθώ σωστός όσον αφορά τους πόρους που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία. Γιατί αν δεν έχει αρκετούς πόρους, τότε θα το βρούμε μπροστά μας και θα συμβεί αυτό κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι στη δικιά μου τη θητεία και θα υπάρξει ένα σκάνδαλο το οποίο θα πλήξει τις δημοσιονομικές αρχές, τις αρχές επί του προπολογισμού. Οπότε από τη μια σας λέω βοηθήστε μας να κρατήσουμε την έκθεση αυτή, να συνεχίζεται κάθε χρόνο. Από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην βρούμε μπροστά μας τις δυσκολίες των περικοπών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Ναι. Τρεις ομιλίες είχαμε ουσιαστικά. Ο λόγος στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Ρούμπικ πρώτος, που είναι η επαφή μας με την ε, ΑΣΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνει η χώρα αυτή τη συνεδρίαση. Ο στόχος είναι να τονίσουμε και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η Acer στην αγορά, εσωτερική αγορά ενέργειας, κυρίως ηλεκτρισμού, να μπορέσει να επιτευχθεί η ενιαία αγορά το ταχύτερο δυνατό. Θέλουμε να καταλύσουμε τα σύνορα και να έχουμε μια ενιαία αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα ΕΦΗ τα ξύπνια δίκτυα θα μπορέσουν μονάχα να λειτουργήσουν αν μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο συνεργασίας μέσα στα πλαίσια και της Acer και των άλλων φορέων. <clears throat> και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι έχετε ανεπαρκής, ανεπαρκές προσωπικό. Θα πρέπει να σκεφτείτε λοιπόν μια καλύτερη διαδικασία συνεργασίας και με τους εθνικούς φορείς ενδεχομένως. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο με απασχολεί είναι το θέμα των ε, τιμολογίων. Υπήρξε μια συζήτηση σε βάθος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, <clears throat> συμφωνήσει ότι δεν θέλουμε να έχουμε χωριστές ζώνες τιμών στα εθνικά σύνορα, γιατί αυτό ουσιαστικά αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και αυτές οι αρχές της ελευθερίας ε, κυκλοφορίας αγαθών και προϊόντων και υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί <clears throat> να δεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν σημαντικό, είναι απαραίτητο να, όταν κοιτάμε να δούμε πού είναι τα προβλήματα αν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή σε μια χώρα, τότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή, την κατάλληλη ικανότητα για παροχή ενεργείας. Προτού λοιπόν καταλήξουμε σε μία απόφαση θα πρέπει να γίνεται αυτή η ανάλυση. Η, ΕΝΣΟΕ, η, συν, Σύνοδος των ε, Ρυθμιστών στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να δίνουν τη γνωμοδότησή τους για τα θέματα αυτά για τον ηλεκτρισμό οι ρυθμιστές, είναι απαραίτητο να γίνεται <clears throat> μια απόφαση με τη συμμετοχή τους. Θα είναι πρόωρο να γίνονται αποφάσεις, να παίρνονται αποφάσεις προτού έχει γίνει ανάλυση από την ΕΝΣΟΕ και την Κομισιόν και ελεγχθούν οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ΕΙΣΕ είναι πολύ σημαντική για το μέλλον, έχει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά θα ήθελα σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη αυτό το οποίο έχει τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχει κατ' επανάληψη αναφέρει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αποφάσεις που γίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αντίστοιχους χώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ συνάδελφο Χάινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πολύ σημαντικό επίσης. Θέλω το σχόλιο σας επί δύο διαφανειών που παρουσιάσατε. Την πέμπτη διαφάνεια η οποία δείχνει τη σύγκληση του κόστους παροχής ε, ε, φυσικού αερίου στην Ευρώπη με τρία διαφορετικά χρώματα, σκούρο γαλάζιο, πιο ανοιχτό σκούρο και μετά ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο στην άλλη διαφάνεια του πώς γίνεται η ρύθμιση εκεί και ο έλεγχος. Το σχόλιο μου αφορά την πρώτη διαφάνεια. Βλέπουμε τις βαλτικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, εδώ έχουμε έναν προμηθευτή, μοναδικό προμηθευτή. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άρα οι τιμές είναι υψηλότερε παρόλο που πιο κοντινή πηγή είναι οι ρωσικές πηγές φυσικού αερίου. Βλέπουμε πολύ συχνά τα στατιστικά στοιχεία αυτού του είδους να έχω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ανταγωνισμός δημιουργεί την αγορά και όχι η κοντινή πηγή. Είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας διατίθεται για να ανοίξουμε τις αγορές. Αυτό είναι το σχόλιο. Ερώτηση τώρα. Η διαφάνεια σελίδα 10. Ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο και ρυθμιζόμενες αγορές. Αυτή είναι φραγμή που δημιουργήσαμε στα κράτη-μέλη μας. Στο φυσικό αέριο, στη Βαλτική, στις Βαλτικές χώρες, Εστονία και Λιθουανία, δεν υπάρχει άλλη πηγή. Είναι φυσικό πρόβλημα που μπορεί να επιληθεί μέσω αγωγών αερίου. Στην περίπτωση της Λετωνίας θα εκπνεύσει ένα εικοσιετές μονοπόλιο που χορηγήθηκε, εγκρίθηκε το 1997. Του χρόνου την άνοιξη θα εκπνεύσει αυτό. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, έχουμε ρύθμιση και στο φυσικό αέριο ή στην ηλεκτρική ενέργεια σε κάτι μελη Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η ρύθμιση των αγορών. Υπάρχει κάποιο φυσικό εμπόδιο και γι' αυτό οι χώρες λένε είναι αδύνατον να μην έχουμε ρυθμιζόμενες αγορές. Αυτό θα ήθελα να καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας. Ο κ. Σταλίτσκα θα μιλήσει τώρα. Και λέει και ο Σταλίτσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την παρουσίαση και την έκθεση. Με τα χαράς να την αναγνώσω προσεκτικά. Βέβαια είναι σέλιδη και χρειάζεται πολύς χρόνος. Και ίσως τα όσα πω τώρα ίσως να φανούν ε, αβάσιμα, διότι ίσως να καλύπτονται αυτά που θα αναφέρω στην έκθεση. Βλέποντας αυτά που έχουμε παραλάβει σε κάθε σελίδα, για κάθε ζήτημα, έχουμε μια σύσταση. Δεν αναφέρει σύσταση, αλλά εμπεριέχεται. Θα εκτιμούσα σαφέστερη ε, διατύπωση. Εθνικές λύσεις για την έλλειψη πόρων και ότι η έλλειψη συντονισμού πολιτικών οδηγεί σε φαύλο κύκλο και δεν είναι αποτελεσματικό σχεδιασμός λέτε. Και λέτε ότι η χρήση μηχανισμό που δώσετε στην αγορά εμποδίζουν την αγορά να ρυθμίσει σωστά την τιμή. Και ο εφοδιασμός ε, σε ηλεκτρισμό είναι κάτι που περιορίζεται αν δεν υπάρχει συντονισμός. Δίνεται μια επιλογή σε κάθε αναγνώστη. Λέτε, δεν εκτιμάται η παρούσα διαθέτηση, αλλά είναι θέμα εθνικό και δεν υπάρχει συντονισμός. Η Acer πρέπει να έχει σαφή θέση. Πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό είναι εις βάρος της αγοράς αυτή η κατάσταση. Καλύτερη θεατύπωση θα ήταν η εξής. Μηχανισμοί δυνατότητες χωρητικότητας είναι τελευταίο ε, μέτρο, αλλά όχι εθνικό μέτρο. Χρειάζεται σαφέστερη γλώσσα όταν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με εμάς τους πολιτικούς. Το περιεχόμενο τώρα είναι σαφές. Η έκθεση είναι καλή. Ίσως να έχω διαφορετική άποψη όσον αφορά το κυτρινόχρωμο τμήμα του χάρτη που αφορά την αγορά φυσικού αερίου. Εκεί αναφερθήκατε σε εύρυθμα λειτουργούσα αγορά. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το καλύψουν περισσότερο, καλύτερα. Φύγοντας σωστά σημεία. Το θέμα των ζωνών τιμολόγηση που ανέφερε ο κύριος Ρούμπικ. Συμφωνώ. Αυτό έχει αντίκτυπο. Όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στις γειτονικές χώρες. Ίσως αν διαβάσω την έκθεση θα μου λυθεί το πρόβλημα. Εν γέννη, όταν είχαμε σχεδιάσει την έκθεση δύο πρωτοβουλία για την ενεργική αγορά, χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο. Έρχεται έγκαιρα αυτή η έκθεση. Ζητήσατε να υπάρχει κατάλληλες, να έχει κατάλληλες δυνατότητες η ε, υπηρεσία σας, η ACE στο μέλλον. Το κατανοούμε. Δεν χρειαζόταν καν να ακούσουμε αυτά που είπε ο Λόρδος Μόγκ. Ποιο είναι το θετικό. Με στευλωμένη αγορά ε, ενεργείας σημαίνει ότι πρέπει να ξανασυδιάσουμε την αγορά. Άρα η Acer μπορεί να παίξει ρόλο. Χωρίς να περιμένει νέες αρμοδιότητες. Αλλά το μέγεθος και η δομή των προβλημάτων θα αλλάξουν, θα εξελιχθούν. Και τότε θα χρειαστεί υποστήριξη η Acer. Το κατανοούμε αυτό. Όταν είχαμε εμείς τη δική μας έκθεση, το αναφέραμε. Συμφωνήσαμε από αυτού. Εγώ θα ήθελα να πούμε το εξής. Πρέπει να δείτε τι σας περιμένει. Όχι το εύρος των προβλημάτων να λυφίσει αυτόν. Άρα ανάλογα με το, με το μέγεθος των προβλημάτων πρέπει να δείτε και ποια είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες τελέχωσης, χρήμα κλπ. που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Προεδρεύων κύριος Κόλιτσεκ. Και τώρα οι απαντήσεις του κυρίου Πότσου και του κυρίου Μόγκ. Έχετε το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία μονάχα θα διεξέλθω αυτό που ελέγχθη για τον Acer και την, τον συντονισμό. Αυτό είναι θέμα για τις Κομισιόν το οποίο η Κομισιόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και ξέρω ότι έχουν κάποιε ιδέε προ την κατεύθυνση αυτή. Ξέρω ότι και αυτοί που ανήκουν στην ΠΕΡΕΚ έχουν και αυτοί τις δικές τους θέσει. Και θα αφήσω το θέμα το οργανωτικό στην Κομισιόν. Έχουμε όμως κάποιους εκπρόσωπους της ΜΠΕΡΕΚ που έχουν και ευθύνη για τα θέματα ενέργειας και υπάρχει κάποια οργανική συνεργασία μαζί τους. Και στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών αναπτύχουμε <clears throat> μια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει σαν στόχο προδραστικά να παροτρύνει την εφαρμογή από τους φορείς που έχουν να κάνουν τα ενεργειακά θέματα, μία εκ, των οποίων είναι η Μπέρεκ. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν κάποια θέματα σε αυτή τη συνεργασία που θα προέλθουν και τα οποία θα ευνοήσουν την πραγματική συνεργασία. Ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ έχω μεγάλη κατανόηση για την γλώσσα που χρησιμοποιείτε και τον στεναρό τρόπο με τον οποίο εσείς ε, λαμβάνετε το λόγο. Όλα αυτά τα οποία λέει η έκθεση όμως αυτή είναι πράγματι έγκυρα. Η έκθεση αυτή μας ε, καταδεικνύει την αναλυτική εγκυρότητα της συζήτησης αυτής για ένα πιο θετικό μήνυμα και εγώ καταλαβαίνω τα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι επειδή τελειώνει η θητεία μου θέλω να φύγω γνωρίζοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια είπα το ίδιο πράγμα, ότι το σύστημα δεν έχει καταρρεύσει ακόμα, δεν έχει γίνει κάποιο σκάνδαλο, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. <clears throat> Για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να έχουμε περισσότερους πόρους με περιορισμένη μοναχά επιτυχία σε ένα θέμα. Δεν ασχολούμαι με τα θέματα του προεπιλογισμού, αλλά αυτό το οποίο γίνεται δεν μπορεί κανείς να το υπερασπιστεί. Ξέρω ότι εσείς είσαστε πιο αισιόδοξοι, αλλά εμεί περιμένουμε ακόμα να δούμε ποιε θα είναι οι προτάσει τη Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει η Κομισιόν όταν αναπτύσσει νέε πολιτικέ θα πρέπει να δίνει και νέου πόρου. Δεν μπορούμε εμεί να αφήσουμε κατά μέρο πόρου για τι νέε προκλήσει και ελπίζω θα υπάρχει και η δυνατότητα να εφαρμόζονται τέλη, ιδίω σε συναλλαγές που έχουν με την οδηγία Δημήτρη για να μπορούμε να δώσουμε περισσότερη χρηματοδότηση στον φορέα μας. Ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τίνει ευήκον ους και θα υποστηρίξει αυτή την ιδέα <clears throat> και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Δυστυχώ αυτό το μήνυμα δεν έχει αποδώσει καρπούς και η ελπίδα μας είναι ότι όπως ε, ελέγχθη η έκθεση αυτή μπορεί να κινδυνεύσει να χαθεί στο μέλλον και αυτό θα είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια. Περιμένουμε ακόμα να δούμε αν θα μας δοθούν οι απαραίτητοι πόροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Πότρετσνίκ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των ζωνών τιμών που έθεσε ο κύριος Ρούμπικ και ο κύριος Ντερίτσκα είναι περίπλοκο τεχνικά η σχέση ανάμεσα στην ενέργεια και την ψηφιακή οικονομία. Με πιο ευφύ δίκτυα χρειάζεται αυτή η σύνδεση. Βέβαια φοβάμαι λίγο, αλλά σίγουρα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, είτε αυτό σημαίνει συνεργασία με την Μπέρεκ, θα δούμε. Εξαρτάται αν η Επιτροπή θα συμφωνήσει, αν θα συμφωνήσει η για συνεργασία μαζί μας. Υπάρχουν πολλές εταιρείες από τις τεχνολογίες πληροφοριών που έρχονται στην ενέργεια και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στον κύριο Κολικάτσικ. Τι πρέπει να γίνει ώστε να αποσύρουμε τις ρυθμισμένες τιμές. Θέλουμε να τις εξαφανίσουμε όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αλλά διατηρώντας κατάλληλη προστασία για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Φυσικά θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός και άρα χρειάζεται δράση και εξελίξεις τόσο σε επίπεδο χοντρικής όσο και λιανικής. Και πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές πηγές φυσικού αερίου σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρισμού ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να επιλέξουν την πηγή και να μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους επιλέγοντας διαφορετικές πηγές. Αλλιώς θα υπήρχε μονοπόλιο στην αρχή. Δεν θέλουμε φραγμούς για την είσοδο στην αγορά λιανικής. Και η τρίτη πτυχή που έχει να κάνει και με τη ρύθμιση αλλά και με τη συμπεριφορά είναι να είναι ενήμεροι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και για τα ωφέλη τα οποία μπορούν να έχουν με την απελευθέρωση. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια λοιπόν, προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με το πρώτο και εν μέρη με το δεύτερο. Να υπάρχουν δηλαδή όσο γίνεται περισσότερες πηγές ενέργειας στην κάθε χώρα. Αυτό είναι το μοντέλο στόχος για μας που το αναπτύξαμε εδώ και μερικά χρόνια εμείς οι ρυθμιστές που έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές όσον αφορά τον προμηθευτή, τον πρώτο προμηθευτή και βέβαια η άρση των εμποδίων. Οι φιλοδοξίες τώρα της σύστασή μας Είπατε ότι θέλετε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, κάπως πιο προδραστικοί. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δείτε την έκθεση, θα βρείτε πολλές ειδικέ συστάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα της ικανότητας της αγοράς είναι ένα περίπλοκο, γιατί δεοδός σε ένα σύστημα χωρίς καμία αποτυχία στην αγορά, χωρίς ε, και να στις τιμές και με περιστήρους καταναλωτές, η αποδοχή των υψηλών τιμών εντάξει, μπορεί να μην χρειάζεσαι αυτό το μηχανισμό, αλλά πρέπει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Στις περισσότερες χώρες τώρα υπάρχει ατέλεια στην αγορά. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο μηχανισμό, capacity mechanism ο οποίος δηλαδή μειώνει στο ελάχιστο τις τρευλώσεις στην αγορά. Και πρέπει να έχουμε και μια περιφερειακή προσέγγιση, ώστε να μην δημιουργήσουμε και εμπόδια μεταξύ των χωρών μελών. Τώρα πρέπει να έρθω στο θέμα των τιμών, της ζώνης τιμών. Ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Μία πτυχή, πάντως, είναι ότι δεν πιστεύω πώς θα εξυπηρετήσει τους καταναλωτές αν μιλάμε για μια αγορά τόσο μεγάλη όσο είναι η ευρωπαϊκή, χωρίς ε, βραχή κυκλώμα. Οπότε, ένας βαθμός μποτελιαρίσματος εμπλοκής είναι κάτι λογικό και στέκει σε ένα τέτοιο σύστημα. Βέβαια, τι κάνεις με τη συμφόρηση αυτή. Μερικές φορές, ακόμα και στην ίδια χώρα μέλος, Σουηδία, Ιταλία, η Νορβηγία, έχει ένα σύστημα εσωτερικών ζωνών, δεν είναι μεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το έχει, προσπαθεί να το ρυθμίσει αυτό με την αγορά και να διασφαλίσει ότι η δυνατότητα που έχει κάθε ζώνη χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πάει πιο μακριά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κάθε τοποθεσία έχει διαφορετική τιμή. Είναι δηλαδή μια διαφορετική ζώνη. Οι ζώνες έγιναν ενία τιμή. Τώρα έχουμε σύνορα που έχουμε κληρονομήσει. Έτσι είναι η πολιτική μας ιστορία αυτή. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο που προσπαθεί να δει τη δομή αυτή των ζωνών έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ζώνες που να μην αντιστοιχούν σε πολιτικά σύνορα αλλά να αντικατοπτρίζουν την ε, πραγματικότητα όσον αφορά τον ηλεκτρισμό στο δίκτυο. Μια καλά σχεδιασμένη αγορά πάντα θα έχει κάποια συμφόρηση και κάποια ικανοποιητική διαχείριση της συμφόρησης αυτής. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Η ερώτηση του κύριου Ρούμπικ δεν ήταν ειδική, αλλά σε συγκεκριμένα σύνορα, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει συμφόρηση. Και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον ρυθμιστή και είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας η αποτελεσματικότητα για την ικανότητα στα σύνορα αυτά και οι διαφορετικές ροές απαιτούν τελικά έναν τέτοιο μηχανισμό απόδοσης ε, ικανότητας. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο γίνεται σωστά. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις να προσθέσω ένα μόνο. Η δικιά μου θέση που ήρθα εδώ να σας τα παρουσιάσω αυτά και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας βασίζεται στη δουλειά που κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στη Λουμπλιάνα και σε όλες τις πρωτεύουσε. και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, τις προσπάθειές τους δηλαδή και το έργο τους. Είναι συλλογικό έργο, όπως είπα και μόνο στη Λουμπλιάνα και αλλού. Και του είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ. Well, thank you much for your Σας ευχαριστώ πολύ για, τις, την παρουσίασή σας. Γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι ιδεώδες. Διακόπτεται το δίκτυο στα πολωνικά και τσεχικά δίκτυα, αλλιώς μπορεί να στευλωθεί το δίκτυό μας από τους ε, ανέμους στη Βόρεια Θάλασσα που φυσούν. Ελπίζω να έχετε δίκιο και στο εγγύς μέλλον όλη η Ευρώπη να είναι κίτρινη. So, ε, Τελικά λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις. Ειδικά την κυρία Ρωμάνα Τζόρνταν, την πρώην συνάδελφό μας, τον κύριο Ποτότσνικ και τον Λόρδο Μόγκ για τη συνεισφορά τους και ελπίζω να προβούμε σε άλλη ανταλλαγή απόψεων τον καινούριο χρόνο. Και εκεί να μας αποδείξετε ότι υπήρξατε επιτυχείς στις προσπάθειές σας. Και για τους συναδέλφους, ήτρε και κολτ κοινή συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο. Έναρξης 9 το πρωί. Εντάφθα, σε αυτή την αίθουσα στο δεύτερο όροφο. Έχετε το υπόψη σας. Θα ψηφίσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ. Γεια σας.